Good Καλημέρα σας, καλημέρα συνάδελφοι. Αρχίζουμε τη συνεδρίαση γιατί είναι φορτωμένη η ημερήσια διάταξη και καλό είναι να μην χάνουμε άλλο χρόνο. Θα προεδρεύσω ε, για ένα τέταρτο περίπου μέχρι να έρθει ο πρόεδρος. Ελάβαμε την πληροφορία ότι χτες η ε, υπήρξε τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία. Η ΕΤΑ στη Γαλλία, η τρομοκρατική βασική οργάνωση, σκότωσε έναν αστυνομικό. Αυτό ήθελα να σας αναγγείλω και θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε. Oh, first Καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κιν Καγκάλ που άρχισε τη συνεδρίαση και άσκησε την Προεδρία όσο εγώ ήμουν απασχολημένος με ένα προηγούμενο θέμα Αρχίζουμε σήμερα. Έχουμε όπως πάντα μία πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη πριν να περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 11 όπως είχαμε αποφασίσει θα ήθελα σήμερα το πρωί να σας πω το εξής. Κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι συμμερίζεται όλοι οι μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να καταδικάσουμε το τρομοκρατικό γεγονός της οποίο συνέβη στη Γαλλία. Δηλαδή τον θάνατο ενός Γάλλου αστυνομικού από τα χέρια της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΤΑ της Βασκικής. όλες οι δολοφονικές απόπειρες, όλες οι τρομοκρατικές ενέργειες κατά της ζωής οποιοδήποτε πολίτη, αυτή την ε, συγκεκριμένη περίπτωση κατά ενός δημοκρατικά εκλεγμένου μέλους της, ε, των διοκτικών αρχών που πολεμούν την δημοκρατία σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε προστατευμένοι. Πρόκειται για άτομα το οποίο προστάτευε τη δική μας ελευθερία. Θα ήθελα λοιπόν όλοι να καταδικάσουμε αυτό το γεγονός. Και είμαι σίγουρος ότι με τον ίδιο τρόπο θα εκφραστεί και ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επόμενη σύνοδο ολομελίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους και ξέρουμε ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές, οι αστυνομικές και όλες οι αρχές είναι κατά αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας. Βεβαίως θέλουμε να εκφράσουμε και την αλληλεγγύη μας προς την οικογένεια του δολοφονηθέντος και αυτό είναι κάτι το οποίο εκφράζουμε προς τις οικογένειες όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ε, στην οικογένειά τους θύματα της τρομοκρατίας. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο σημείο της ημερήσιας διάταξης που ανήγγειλε η συνάδελφος Κιν Καγκάλ. Πρόκειται για το Σημείο 11 τη ημερησία, δηλαδή την έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση τη Επιτροπή. Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Έχουμε να κάνουμε εδώ με μία γνωμοδότηση, η συντάκτρια της ε, γνωμοδότησης, του σχεδίου γνωμοδότησης, είναι παρούσα. Η έκθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι ακόμη στη διάθεσή μας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας προτείνω να προτείνουμε μια κατάθεση τροπολογιών το τέλος της παρούσης εβδομάδας, 19 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι, ώστε να μπορέσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης να το ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδριασή μας, στις 7 Απριλίου δηλαδή. Θα ακούσουμε τώρα την εισηγήτριά μας, την κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, έχετε το λόγο. Good morning, Mr. President. Uh, good morning, everybody. Καλημέρα, κυρίες και... Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Ε, και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να εκφράσω την συμπαράστασή μου και τα συλληπιτήριά μου. Η πρόταση για κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών είναι πολύ επίκαιρη τα τελευταία χρόνια αλλά και φέτος Είχαμε σοβαρές φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη και, στο εξωτερικό, και εκτός Ευρώπης. Στην τελευταία ολομέλεια του Στρασβούρου υιοθετήσαμε ψήφισμα για τις ε, μεγάλες καταστροφές στην Μαδέρα ε, και ε, στην Ευρώπη. Θέλουμε ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση καταστροφών. Το ε, η έμφαση στο ε, έγγραφο της Κομισιόν επικεντρώνεται στην ε, αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών. Τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών δίνουμε έμφαση στην ανάγκη προστασίας των πολιτικών ελευθεριών και δράσης μετριασμού των επιπτώσεων αυτών των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Έτσι λοιπόν στο σχέδιο ε, προτείνω ε, σχέδιο γνωμοδότησης. Δυστυχώς το σχέδιο γνωμοδότησης διετέθη στα μέλη μόλις τώρα, χθε το απόγευμα συγκεκριμένα, και δεν υπάρχει σε όλες τις γλώσσες. Προτείνω λοιπόν κύριε Πρόεδρε, αντί να προβλέψουμε τη 19η Μαρτίου για την προθεσμία, αν είναι δυνατόν να μετατεθεί μέχρι τις 12 Απριλίου η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών λαμβάνοντας υπόψη ότι η, έκθεση, η ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ θα γίνει ή 3 ή 4 Μαΐου. Άρα υπάρχει αρκετός χρόνος για τις τροπολογίες και έτσι θα ασκήσουν όλα τα μέλη της Επιτροπής στο δημοκρατικό τους δικαίωμα να υποβάλουν προτάσεις για να βελτιώσουν τη γνωμοδότησή μου. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Φερέιρα είναι μια καλή έκθεση και επιπροσθέτω, στο σχέδιο γνωμοδότησης μου εξ ονόματος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ προσέθεσα μια σειρά προτάσεων που θα ήθελα εν συντομία να παρουσιάσω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ίσως κάποιοι δεν την έχουν διαβάσει. Κάποιες προτάσεις είναι οι εξής. Η πρώτη χαιρετίζει την αυξανόμενη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανάπτυξη των πολιτικών ασφάλειας μετά την ε, θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, χρειάζονται διαβουλεύσεις σε όλα τα στάδια. Ε, ε, υπογραμμίζω με την σημασία των πολιτικών συζητήσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και διαφορών εμπλεκομένων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων μελών της κοινωνίας των πολιτών. Τρίτον, υπογραμμίζομαι ότι η αρχή της μη διάκρισης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, να συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις. Ε, επίσης θέλουμε αποτελεσματική παρακολούθηση των ε, προσπαθειών ανακούφισης ώστε να ε, γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα συμπεριλαμβάνοντας προληπτικές δράσεις όπως την αντιμετώπιση ε, κλιματικής συμπεριφοράς, εμπορίας ανθρώπων κλπ. Ε, τέλος, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετεί στρατηγικές που θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου ε, στις περιβαλλοντικές κρίσεις από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Καλούμε την Κομισιόν να θέσει σαφείς προτεραιότητες για την παροχή υποστήριξης στις χώρες που επλήγησαν από την καταστροφή. Δηλαδή, διατάξεις που θα προβλέπουν ε, τον χώρο όπου θα στεγάζονται οι πληγέντες, ε, υγειονομικές υποδομές κλπ. Τέλος, θέλουμε συστήματα έγκαιρης ε, προειδοποίησης και προγράμματα για την γενικότερη ενημέρωση. Θέλουμε επίσης να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο καταστροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ χρειάζεται ε, γενικότερη συλλογή πληροφοριών και ενημέρωση σε σχέση με τους κινδύνους και το κόστος των καταστροφών σε επίπεδο ενωσιακό. Επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας οριζόντιος συντονισμός, μηχανισμός συντονισμού. Ε, επίσης αναφέρομαι στον ε, ρόλο της μόνιμης επιτροπής για την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική ασφάλεια η οποία θεσπίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου ε, του 2010 από τους 27 ε, υπουργούς ε, ΔΕΗ στις Βρυξέλλες για αποτελεσματικό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των αρχών διαχείρισης των συνόρων. Τέλος, συνιστούμε την θέσπιση ε, ενός χρηματοδοτικού μέσου ειδικού για την πρόληψη καταστροφών που θα συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες ε, προστασίας κυρίως ανθρώπων αλλά και του περιβάλλοντος και της περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ε, δεν χρειάζεται βέβαια να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι συμφωνούμε απόλυτα με την δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου πιο ευέλικτου και ισχυρού ένα μέτρο το οποίο υπογραμμίζεται ε, σαφώς και από τον εισηγητή της Επιτροπής ΕΝΒΗ οι επεπλεγμένες διαδικασίες ε, που πρέπει να ακολουθήσουν οι χώρες για τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης που έχει ετήσιο προϋπολογισμό 1 δις ευρώ ε, αφήνει την, ε, δεν αφήνει άλλη επιλογή στην Επιτροπή και την Ισπανική Προεδρία από το να ενεργοποιήσει την ε, αναθεώρηση του κανονισμού για το Ταμείο Λιλεγγύης. Ένα τελευταίο σημείο είναι ότι τώρα που η Ευρώπη έχει τη μοναδική ευκαιρία να διαμορφώσει την νέα εξωτερική, υπηρεσία εξωτερικής δράσης για μια ολιστική και συνεκτική πολιτική, ε, εξωτερική πολιτική, αλλά και πολιτική ασφάλειας, όχι μόνο ε, μεταξύ των 27, αλλά και στις τρίτες χώρες, νομίζω ότι είναι καιρός να έχουμε αυτή την ενωσιακή προσέγγιση για τη διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών ως μια προτεραιότητα. Και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ε, όταν θα συζητήσουμε ε, για το ε, χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας ε, να ακούσω τις προτάσεις και συστάσεις σας. Thank you, Mrs. Let's hear maybe some comment from... Κυρία Παπαδοπούλου, θέλει η Κομισιόν να κάνει κάποιο σχόλιο. Πρώτα απ' όλα δεν βλέπω κανένα εκπρόσωπο από το Συμβούλιο παρόντα. Ναι, ναι, κάποιο είναι εδώ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελε η Επιτροπή να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την ε, συνεισφορά της στην έκθεση του κυρίου Φεραίρα για την ε, κοινωτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Προσπαθούμε να έχουμε ισοσκελισμένη προσέγγιση και στον τρόπο με τον οποίο το αποκρινόμεθα και προσπαθούμε κυρίως να ε, ασχοληθούμε και με την πρόληψη και την αλληλεγγύη πριν από αυτή την ανακοίνωση είχαμε θέσει κίνηση, διάφορες πρωτοβουλίες, τις βέλτιστες πρακτικές, την ανάλυση κινδύνου, την ε, γνώση των ε, διαφόρων καταστροφών και θέλουμε να μελετήσουμε και τον τρόπο της καλύτερης ε, ένταξης της πρόληψης στα δημοσιονομικά μέσα τα οποία διαθέτουμε για την προστασία ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Η κυρία Σεσίλια Βίγκστρομ ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την πολύ ισορροπημένη έκθεση που μας παρουσίασε. Εάν Ήδη η ανακοίνηση ε, της Επιτροπής πιστεύω ότι είναι μια καλή ανακοίνωση και έχοντας ακούσει και την εισηγητρία μπορούμε να πούμε ότι σήμερα οι κοινωνίες όλες μας είναι πάρα πολύ ευάλωτες εξαιτίας των καταστροφών. Των καταστροφών οι οποίες πολλές φορές ήταν και ανθρωπογενείς και οφείλονταν σε κακή θέληση κάποιων αλλά και φυσικές καταστροφές. Ας υπενθυμίσουμε το τσουνάμι, την ε, καταστροφικό σεισμό της Αιτής. Σήμερα λοιπόν είναι περισσότερο σαφές από ποτέ ότι ο άνθρωπος μπορεί να προκαλέσει πολλές καταστροφές ε, επίσης. Ε, ακούμε τι γίνεται με τις τρομοκρατικές ε, ενέργειες, πόσα θύματα υπάρχουν. Βλέπουμε πόσο η αστυνομία πρέπει πάντα να προστατεύει όλους όσοι ζουν στις ε, ελεύθερες, στις ε, ανοιχτές κοινωνίες τις σημερινές. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό σήμερα και επίκαιρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παπαδοπούλου, διότι με την έκθεσή της κάνει έκκληση να υπάρχει συνεργασία, συνεργασία με όλη την ε, κοινωνία των πολιτών, να μην υπάρχουν διακρίσεις, ενώ συγχρόνως τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα να γίνονται σεβαστά παντού. Πιστεύω ότι μετά από οποιαδήποτε ε, καταστροφή τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται πραγματικά εν κινδύνο. Πρόκειται για καταστάσεις πολύ ευάλωτες. Βεβαίως δεν είναι όλες οι καταστάσεις ίδιες και ε, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου. Υπάρχουν ε, οικολογικές καταστροφές στην Νότια Ευρώπη όπως οι διάφορες ε, ε, πυρκαγιές από τις οποίες υπέφερε η Ελλάδα εδώ και χρόνια που πραγματικά είναι οικολογικές καταστροφές. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλούμε για τέτοιου είδους θέματα και να μην ξεχνάμε ότι και σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμβούν καταστροφές. Η στρατηγική μας θα πρέπει να βασίζεται όπως γίνεται στην ε, Νότια Ευρώπη, οι διάφορες περιφέρειες, οι περιοχές να είναι υπεύθυνε για την πρόληψη τέτοιου είδους καταστροφών. Δεν υπάρχει όμως τέτοιου είδους σύστημα παντού. Εμείς στις βόρειες χώρες έχουμε χειμώνες για μήνες. Δεν υποφέρουμε από μεγάλες ζέστες, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα μέσα υποδομής τα οποία διαθέτουμε για να προστατεύουμε όλες τις περιοχές μας. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι όταν κανείς είναι μόνος του για να αντιμετωπίσει μια καταστροφή είναι μόνος του, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αλληλεγγύη. Αναφέρεται στην ε, έκθεση ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο. Εάν δεν μπορούμε να κάνουμε μια αποτελεσματική νέα οργάνωση, καλύτερα να ενισχύσουμε τους ήδη υπάρχοντες ε, οργανισμούς. Ας κάνουμε πιο ανταγωνιστικές τις οργανώσεις που έχουμε, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουμε νέες γραφειοκρατικές δόμεν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις ε, καταστροφές που αντιμετωπίζει πότε ο Βορράς, πότε ο Νότος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ενισχύσουμε πριν να δημιουργήσουμε νέους οργανισμούς αυτούς που ήδη υπάρχουν. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Γκυλιόμ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν είναι άμεσα για το θέμα της κυρίας Παπαδοπούλου. Άκουσα να γίνεται μια από συναδέλφους για την καταδίκη ενός χτυπήματος του ΕΤΑ στη Γαλλία. Ήθελα να πω μόνο δύο λόγια γι' αυτό. Φυσικά όλοι μας είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να καταδικάζεται η τρομοκρατία πάσης μορφής και βία πάσης μορφής αλλά λίγο μέτρο αυτή τη στιγμή διότι από ό,τι ξέρω είμαστε στη φάση της έρευνας η ανάκριση που ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα του ΕΤΑ από ό,τι ακούω εγώ. Χθε έγινε αυτό. Γάλλοι αστυνομικοί κλήθησαν ε, για μια κλοπή αυτοκινήτου τελικά ξελίχθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών ένας από τους τέσσερις ανήκει στον ΕΤΑ από αυτούς που ενεπλάκησαν, αλλά δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια κατά της γαλλικής αστυνομίας εκ μέρους του ΕΤΑ. Εγώ δεν είμαι ούτε μέλος των μυστικών υπηρεσιών της γαλλικής αστυνομίας, ούτε αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε προεκλογική καμπάνια στη Γαλλία και θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια ορισμένοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν ποινικά δικήματα στη φάση της προεκλογικής καμπάνιας. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο και τώρα. Φυσικά και επαναλαμβάνω, καταδικάζω οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ας περιμένουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Διαζεμέρα. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες συμπληρωματικές προφορίες, Σίλβη. Ε, ο κρατούμενος λέγεται Χωσέβα Φερνάντο Ατούρες και όταν τον ε, ε, συνέλαβε η Γαλλική Αστυνομία είπε ότι είναι μέλος της ΕΤΑ. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τρομοκρατική πράξη με απόπειρα της ΕΤΑ και όπως είπατε και εσείς και είπε ο Πρόεδρος, θα πρέπει με απόλυτη σαφήνεια να καταδικάξουμε αυτή την δολοφονική πράξη. Any Πρόεδρος, θέλει κανείς άλλο το λόγο. Παρακαλώ όμως να είμαστε στο θέμα μας. Το σημείο 11 της της διάταξης. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Σωστό, σωστό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο κυρία Παπαδοπούλου για την γνωμοδότησή της. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό που έχει και διαφορετική προοπτική. Εσεί, γράψατε στην γνωμοδότησή σας ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, διαβίας μετανάστευση. Συμφωνώ. Αυτό το θέμα των φυγάδων λόγω κλιματολογικών συνθήκων είτε μέσα στην Ένωση είτε εκτός Ένωσης φυγάδες, πρόσφυγες, θα αυξηθεί σιγά σιγά με τον χρόνο και η Επιτροπή Ελευθεριών σωστά στρέφει την προσοχή της στο θέμα αυτό. Χθες συζητήσαμε το πλήρες πακέτο για το άσυλο. Θα το συνεχίσουμε αυτό και στους επόμενους μήνες. Επίσης θα συζητηθεί για το Δουβλίνο, για θέματα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών για την αποδοχή προσφύγων. Πολλοί πρόσφυγες προς την Ευρώπη ήδη προέρχονται από καταστάσεις ε, βίας που με τη σειρά του μπορεί να έχουν δημιουργηθεί και από πλημμύρες, ε, ξηρασία κλπ. ή ανθρωπογενείς καταστροφές είτε φυσικές καταστροφές. Όλο αυτό μας δείχνει ότι πρέπει να φροντίσουμε τους πρόσφυγες που ήταν υποχρεωμένοι να φύγουν και για λόγους κλιματολογικούς. Και παρακαλώ την κυρία Παπαδοπούλου αν θα ήθελε να σκεφτεί και το θέμα αυτό και ενδεχομένως να το συμπεριλάβει στην έκθεσή της. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπόνς. Κύριε Πρόεδρε, Όπως ε, είπαν και οι συνάδελφοι, μιλάμε για ένα θέμα ανθρωπογενών καταστροφών στο κλίμα. Μιλήσαμε και για τρομοκρατικές ενέργειες, όλα τα ρίξαμε σε ένα σακί. Αυτό δεν έχει νόημα. Η επίθεση που έγινε στο Παρίσι είναι καταδικαστέα. Ωστόσο, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει αυτό με τη συζήτηση που κάνουμε για τις ανθρωπογενείς καταστροφές. Η άνηση μεταχείριση τι σχέση με τις ανθρωπογενείς καταστροφές και γιατί να κατηγορούμε τους ανθρώπους για τις αλλαγές στο κλίμα. Γιατί, όπως μας είπε και η IPCC, έχει γίνει μαγείρεμα των αριθμών. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μπει λίγο τάξη στη συζήτησή μας. Εδώ συζητάμε για θεομηνίες, φυσικές καταστροφές. Η γνώμη μου είναι ότι όταν συζητάμε για φυσικές καταστροφές υπάρχουν ε, ταμεία έκτακτης ανάγκης δεν έχει σχέση αυτό με την Ένωση να έχουμε αυτό το υπερκράτος στην εδώ που δεν το θέλουμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ των πραγμάτων που συζητάμε είναι γελίος ο τρόπος με τον οποίο συζητήσαμε μέχρι τώρα σήμερα το πρωί όλα αυτά τα θέματα μαζί Πρόεδρος μετά από τη συζήτηση αυτή σημειώνουμε την πρόταση της κυρίας Παπαδοπούλου να οριστεί 12 Απριλίου προθεσμία για τις τροπολογίες για να ψηφίσουμε αρχές Μαΐου Yes, yes, yes. We're voting in Στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε. τον Απρίλιο και το Μάιο Ολομέλεια. Σημειώστε το αυτό. 12 Απριλίου τροπολογίες. Περνάμε στο 12. Δικαίωμα διερμηνίας και μετάφρασης σε ποινικές διαδικασίες. Έχουμε μια πρωτοβουλία που συζητήθηκε αρκετά Ζητάμε ένα νομικό εργαλείο σε θέματα διαδικασίας και τα δικαιώματα που τα σχετικά. Στην πρώτη προσπάθεια της Κομισιόν δεν απέδωσε γιατί τα κράτη-μέλη δεν συμφώνησαν με την πρόταση για την απόφαση πλαίσιο του 2004. Δεύτερη προσπάθεια του 2009 όπου η Κομισιόν έκανε νέα πρόταση για απόφαση πλαίσιο για το δικαίωμα διερμηνίας και μετάφρασης σε ποινικέ διαδικασίες. Οι προσπάθειες της Ειδικής Προεδρίας απέδωσαν καρπούς και το Σχετικό Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου κατέληξε σε συμφωνία σε ένα πακέτο για τρία έγγραφα Πρώτον, ένα ψήφισμα του Συμβουλίου για roadmap για την ενίσχυση των δικαιωμάτων ε, υπόπτων ή κατηγορούμενων σε ποινική δίκη. Ένα σχέδιο απόφαση πλαισίου του Συμβουλίου για το δικαίωμα μετάφραση διερμηνία σε ποινικέ διαδικασίε προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα τη διαδικασία υπόπτων ή κατηγορουμένων. Και τρίτο, ψήφισμα του Συμβουλίου που ενισχύει την εφαρμογή από τα κρατημέλη του δικαιώματο διερμηνίας και μετάφρασης σε ποινικέ διαδικασίες. Άρχισε να ισχύει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Αυτή η δεύτερη προσπάθεια με το νομικό αυτό εργαλείο δεν λειτουργήσε και η απόφαση πλαίσιο και το ψήφισμα δεν εγκρίθηκαν τυπικά. Κατά συνέπεια, 13 μετά μάλλον 13 χώρε χώρες μέλη αποφάσισαν να μια πρωτοβουλία για οδηγία για τα δικαιώματα διερμηνίας μετάφρασης. Στο περιεχόμενο ήταν το ψήφισμα του Συμβουλίου για την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη του δικαιώματος διερμηνίας και μετάφρασης ποινικέ διαδικασίας ε, είναι προσθετημένο στο σχέδιο πλαισίου απόφαση, αλλά δεν είχε μπει στο κείμενο τη πρόταση για οδηγία από τα κράτη-μέλη, η εισηγήτρια ζήτησε τη Συμβουλή των Νομικών Υπηρεσιών του Κοινοβουλίου κατά πόσον το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει ένα τέτοιο ψήφισμα ή οτιδήποτε άλλο μη δεσμευτικό νομικό εργαλείο υπό το νομικό πλαίσιο της συνθήκη της Λισαβόνας και τη δυνατότητα να μπει το περιεχόμενο του σχεδίου ψηφίσματος στις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας. Παράλληλα, η Κομισιόν αποφάσισε να υποβάλει μια πρόταση στο ίδιο θέμα και με ευχαρίστηση θα ακούσουμε την παρουσίαση αυτής της νέας πρότασης. Καταρχήν, το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Σάρα Λούτφορτ, και μετά οι νομικές υπηρεσίες και μετά η Κομισιόν. Κυρία Ράντφορντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, θα κατάλαβαν οι συνάδελφοι από την εισαγωγή, είχα μεγάλη περίοδο κυκλοφορίας, έξι χρόνια κυοφορία. Πάντως, πιστεύω ότι πλησιάζουμε σε αίσιο πέρας. μεταξύ του 2004 και του 2007 έγινε μια προσπάθεια για συμφωνία σε ευραία μέτρα για πολλά δικαιώματα επί της διαδικασίας. Φυσικά όλα αυτά τα υποστήριξε το Κοινοβούλιο, αλλά το 2007 οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν πουθενά. Πέρυσι η Σουηδική Προεδρία ξανάφερε στη ζωή τη συζήτηση με μια βαθμία διαδικασία μέτρων προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα νομικό εργαλείο Βέβαια μπορούμε να δούμε το ποτήρι μισό άδειο ή μισό Εξαρτάται. Εγώ θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Αυτός ο δικός χάρτης εγκρίθηκε τον Οκτώβριο με βάση το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και όπως είπε και ο Πρόεδρος τον Ιούλιο η Κομισιόν έκανε πρόταση για το πρώτο μέτρο του roadmap έκανα ένα ε, σχέδιο έκθεσης για την απόφαση πλαίσιο συζητήθηκε στην Επιτροπή μας τον Νοέμβριο οι συνάδελφοι την υποστήριξαν μετά άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας στο μεταξύ εννοώ μας μπέρδεψε κάπως το συζήτησα με την Κομισιόν κατά πόσο γρήγορα μπορούσε να μας κάνει μια πρόταση για οδηγία που είναι το νέο εργαλείο της συνθήκης της Λισαβόνας. Βέβαια είχαμε μεταβατική περίοδο, τέλος της εντολής της Κομισιόν. Ο πρόεδρος Μπαρόσο θεώρησε ότι καλό θα ήταν να μην κίνηθει κάτω από αυτές τις συνθήκες και χάσαμε μερικούς μήνες. Αρχικά εγώ το είχα προτείνει. Τα κράτη-μέλη να πάρουν πρωτοβουλία. Δεν ε, είμαι πάντα υπέρ των πρωτοβουλειών των κρατών μελών, διότι συχνά είναι πρωτοβουλίες press conference στην αρχή της κάθε προεδρίας. Έρχεται ο Υπουργό Ιστορικών, ο Υπουργό Υπεύθυνο για τη Μετανάστευση, κάποιος άλλο υπουργός Κάνουν προτάσεις που δεν είναι και πολύ χρήσιμες. Ωστόσο, αυτή η περίπτωση είναι διαφορετική. Ήταν μια ρεαλιστική λύση. Και τελικά 13 χώρες μέλη υπέγραψαν το κείμενο αυτό της πρότασης. Η έκθεσή μου στηρίζεται σε αυτή ακριβώς την πρωτοβουλία των κρατών μελών. Αυτά το Δεκέμβριο, άρθρο 76 της Συνθήκης. Και μετά οριστικοποιήθηκε η εκθεσή μου και την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν έκανε την πρότασή της. Τότε στηριστήκαμε στο κείμενο του, συνο... του Συμβουλίου, δεν σημαίνει ότι είμαι ικανοποιημένη με το κείμενο αυτό, κάθε άλλο. Τα κράτη-μέλη το ενέκριναν ως κείμενο μια συμφωνία μεταξύ τους βάσει βάση το σχέδιο ε, απόφασης πλαισίου του 2009 με βάση την ομοφωνία. Βέβαια η ομοφωνία ε, κινείται στο επίπεδο ελάχιστου κοινού παρονομαστή όσον αφορά τις φιλοδοξίες. Αναπόφευκτα υπέβαλα μερικές ε, πολύ έντονου ύφους τροπολογίες για να βελτιωθεί το κείμενο σε τρεις βασικούς τομείς. Πρώτον, διερμηνία για επικοινωνία με τους δικηγόρους, με τον δικηγόρο του υπόπτου, από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Στην ανάκριση, στο, στην ανάκριση στην αστυνομία και στη διάρκεια της δίκης. Στην ακροματική διαδικασία. θεωρώ αναγκαίο για να υπάρχει δικαιοσύνη και να μπορεί ο κατηγορούμενος να καταλαβαίνει τι λέγεται. Το κείμενο της Κομισιόν με καλύπτει στο σημείο αυτό. Δεύτερο, πεδίο τροπολογιών, οι γραπτές μεταφράσεις θα πρέπει να γίνονται για όλα τα βασικά κείμενα η κατηγορία, το κατηγορητήριο, ε, το ένταλμα σύλληψης κλπ. Ενώ το άλλο κείμενο λέει προφορικές συνόψεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Εγώ δεν αποκλείω τις προφορικές συνόψεις όπως κάνει η Κομισιόν, αλλά ζητάω αυστηρά κριτήρια. Όχι μόνο την παρουσία του δικηγόρου, του κατηγορούμενου, αλλά υπάρχουν πρακτικά όταν έχουμε προφορικές συνόψεις. Να ξέρουμε τι υπόθηκε στον ύποπτο. Τρίτο, οι όροι κάτω από τους οποίους μπορεί ο ύποπτος να πει δεν το θέλω το δικαίωμα αυτό. Δηλαδή, πριν δοθεί αυτή η απαλλαγή, να έχει νομική συμβουλή και η εντολή αυτή να δοθεί γραπτά να είναι σαφής και να μην είναι κατά του δημοσίου συμφέροντος. Εδώ πάω πιο πέρα από το κείμενο της Κομισιόν. Αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα. Υπάρχουν κι άλλα ελάσσονα. Μας χάρη ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης, όπως επίσης και η Ευρωπαϊκή Συνθήκη, η εφαρμοσιμότητα αυτών των γλωσσικών δικαιωμάτων να ξεκινάει όχι μόνο όταν γίνεται μια ανάκριση, αλλά και από τη στιγμή που ο ύποπτο γνωρίζει τι είδους υποψία τον βαρύνει. Και όχι απλώ να πληροφορηθεί ο ύποπτο ότι τον βαρύνει η υποψία. Το δικαίωμα πρέπει να καλύπτει όλες τις φάσεις της διαδικασίας από την αρχή μέχρι το τέλος. Άρα και μετά την καταδίκη. Στη χώρα μου μπορείς να καταδικαστείς και μετά να υπάρξουν εκθέσεις κλπ. Πριν βγει η τελική απόφαση. Αυτό εξακολουθεί να είναι κομμάτι της ποινική διαδικασίας. Να έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες έφεσης. Τότε λύγει το θέμα. Επίσης γραπτά πρέπει να γνωστοποιούνται τα δικαιώματα στον ύποπτο τα δικαιώματα που έχει διερμηνή και μετάφραση. να καλύπτονται άτομα τα οποία έχουν αναπηρία, η έφεση να γίνεται σε δικαστική αρχή, να πρέπει να οριστεί ο μηχανισμός έφεσης, να υπάρχουν όροι για την εκπαίδευση και ε, προσόντα προκειμένου να καταγραφεί κάποιος ως διερμηνέας και μεταφραστής για την περίπτωση αυτή χρήση οπτικοακουστικών μέσων καταγραφής, κατάλληλοι χώροι, προθεσμίες, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανάγκη σε διερμηνία και μετάφραση κλπ. Αυτές είναι ελάσσονες τροπολογίες. Μετά έχουμε το θέμα πώς στην οδηγία θα μπει θα μπουν οι όροι που βάλανε τα κρατη στο ψήφισμα. Η νομική μας υπηρεσιά μας λέει ότι τα κρατη δεν μπορούν να εγκρίνουν ταυτόχρονα ψήφισμα αν εγκρίνουν οδηγία. Με βάση τη νέα συνθήκη μπορούμε στην οδηγία να βάλουμε μέτρα πάνω χάρη για την κατάρτιση των δικαστών, ότι υπάρχει νομική βάση γι' αυτό. διαδικαστικά πρότεινα να κρατηθούμε στην πρωτοβουλία των κρατών μελών. Η έκθεση να στηριχθεί μόνο σε αυτό. Οτιδήποτε άλλο. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θα περιπλέξει τα πράγματα, θα τα καθυστερήσει. Και χρήσιμο είναι να εμπνευστούμε μεν από το κείμενο της Κομισιόν αλλά όχι διαδικαστικά να στηρίξουμε την έκθεσή μας στο κείμενο της Κομισιόν. Γιατί προσπαθώ να ισορροπήσω με μία έκθεση μεταξύ δύο άλλων κειμένων και μου είναι δύσκολο να το πετύχω αυτό. Τίποτα βέβαια δεν μας εμποδίζει να δούμε την διατύπωση του κειμένου της Κομισιόν και να εμπνευστούμε. Αυτά είχα να σας πω κύριε Πρόεδρε. Στη διάθεση του συνδέφου να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Ζήτησα από τους κοιόδες εισηγητές μια στενή προθεσμία μέχρι την Τρίτη την επόμενη εβδομάδα, 23 του μηνός. 12 η ώρα, προθεσμία τροπολογιών. Ξέρω ότι δεν είναι μακριά η επόμενη Τρίτη και το κείμενο το έχουμε μόνο σε τρεις γλώσσες. Αγγλικά, Ισπανικά, Ρουμανικά. Την Παρασκευή θα το έχουμε σε όλες τις γλώσσες. Αν οι το δέχονται αυτό, θα είναι χρήσιμο, γιατί μετά έχουμε το Πάσχα και θα έχουμε καθυστέρηση. Εγώ θα ήθελα να μπορούμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 7 Απριλίου προς Ανατολισμός και να περάσουμε στην Ολομέγεια το Μάιο ή το αργότερο Ιούνιο. Αν συνάδελφοι συμφωνήσουν, θα μου είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ευχαριστώ κυρία Λάντφορντ. Και τώρα η Προεδρία, πριν από την Προεδρία και την Κομισιόν, καλό είναι να ακούσουμε τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. παρακαλώ, εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας, ο προσκεκλημένος μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε την νομική μας ε, γνωμοδότηση σχετικά με την προτινόμενη οδηγία για τα δικαιώματα διερμηνίας και μετάφρασης σε ποινικέ διαδικασίες. Ειδικότερα ζητήσατε από την νομική υπηρεσία να αναλύσει αν το Συμβούλιο μπορεί να υιοθετήσει ένα ψήφισμα όταν ε, εξετάζει σχέδιο οδηγίας στον ίδιο τομέα. Δεύτερον, αν το προτινόμενο ψήφισμα μπορεί να εγκριθεί ως σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 292 ε, της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν το περιεχόμενο του σχεδίου ψηφίσματος μπορεί να ενταχθεί στις αιτιολογικές σκέψεις της προτινόμενης οδηγίας. Για να συνοψίσω τη γνωμοδότησή μας επί των δύο ε, ερωτήσεων Καταλήγουμε ότι όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 296 της Συνθήκης, όταν εξετάζομαι την προτινόμενη οδηγία για τα δικαιώματα διερμηνίας και μετάφραση σε ποινικές διαδικασίες, επί τη βάση του άρθρου 82.2 της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, είναι υποχρεωμένα να απόσχουν από την έγκριση πράξεων που δεν προβλέπονται ε, στον τομέα που καλύπτει το άρθρο 82. Αυτό το άρθρο δεν προβλέπει την έγκριση ούτε ψηφισμάτων του Συμβουλίου και των κυβερνήσεων των κρατών μελών, ούτε συστάσεις του Συμβουλίου. Ε, ακόμα και αν το άρθρο 292 της ε, συνθήκης παρέχει στο Συμβούλιο γενικό δικαίωμα έγκρισης συστάσεων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 296 δεν προβλέπεται αυτή. Ε, προβλέπει πιο συγκεκριμένη διάταξη στις ε, παρούσες συνθήκες. Ε, αναφέρθηκε ότι η γνωμοδότησή μας είναι πολύ περιοριστική και ότι ο πραγματικός λόγος ύπαρξης του 296-3 είναι να ε, προλάβει να αντικαταστήσουν ένα μέσον με ένα άλλο τα θεσμικά όργανα. Αν είναι αυτός ο λόγος ύπαρξης διάταξης, δεν είναι, δεν είναι λόγος, αν η συνθήκη προβλέπει ότι μόνο μια οδηγία μπορεί να εγκριθεί, τότε η υποκατάσταση κανονισμού θα είναι παραβίαση της συνθήκης με ή χωρίς το άρθρο 296 της ΛΕ. Έτσι, η νομική υπηρεσία θεωρεί ότι ο νομοθέτης θα πρέπει να απόσχει από την υιοθέτηση ε, ψηφίσεων και συστάσεων στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας για την οδηγία που προτείνεται. Σε ό,τι αφορά το τρίτο ερώτημα, θέλουμε να πούμε ότι ο λόγος του προημίου σε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι να υποδηλώσει τους λόγους για τις διατάξεις επί της ουσίας. Όπως αναφέρθηκε και από το 10, οι λόγοι πράξης νομοθετικού περιεχομένου επιτρέπουν σε, στον ενδιαφερόμενο να ε, βεβαιωθεί για τις συνθήκες ε, στα πλαίσια των οποίων άσκησε το θεσμικό όργανο της εξουσίας τους. Ε, ε, συμπερίληψη ε, μη νομοθετικών διατάξεων όπως αυτές που αναφέρονται στο σχέδιο ψηφίσματος ε, αντιβαίνουν και στο άρθρο 296 και στην ομολογία που αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε τώρα πρώτα την Προεδρία και μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Αγγιλέρα, παρακαλώ. Sí, muchas gracias, señor presidente, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την δυνατότητα να σας παρουσιάσω τη θέση της Προεδρίας σε αυτό το θέμα. Θα ήθελε η Προεδρία πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την έκθεσή της και να σας πει ότι το Συμβούλιο είναι στην διάθεσή σας για να μπορέσει να καταλήξει σύντομα σε ικανοποιητική και ταχεία συμφωνία για όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε κάποια στοιχεία που προϋπήρχαν πριν την έκθεση και να τα έχουμε κατά νου για να είμαστε σίγουροι ότι θα προχωρήσουμε προς ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την εναρμόνιση όλων των ε, διαδικασιών, πράγμα το οποίο επιθυμούμε όλοι να ολοκληρωθεί. Αυτό θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος και θα βοηθήσει και κάποια επόμενα βήματα να ολοκληρωθούν. Αυτή είναι έννοια λοιπόν, όπως λέγω, το Συμβούλιο, η Προεδρία είναι στην απόλυστη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η έκθεση της εισηγήτριας και μπορεί να μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό. Γνωρίζουμε ποια είναι τα θέματα τα οποία τίθενται επιτάπητος προς συζήτηση. Ξέρετε ποια είναι τα θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής, τι απασχολεί τα κράτη-μέλη και η διάθεσή μας είναι να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συμφωνία για την έκθεση αυτή στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης. Όπως ξέρετε πρέπει να υπάρξει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από διαπραγμάτευση μαζί σας. Ήδη στο Συμβούλιο έχουν αρχίσει επί αυτού του θέματος οι πρώτες συζητήσεις βάσει των πρώτων τροπολογιών που καταθέσατε και έχουμε λάβει και είμαστε στην ε, απόλυτη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε και να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να καταλήξουμε, επαναλαμβάνω, το συντομότερο δυνατό σε συμφωνία. Και βεβαίω θέλουμε να συνεργαστούμε όχι μόνο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει να είναι παρούσα και να συμμετέχει ενεργά σε όλε τι συζητήσει. Αυτή είναι η δική μα απόψη. Θα θέλαμε επίση να πούμε ότι μας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύστοχο το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η συγγήτρια, διότι μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις και να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι λοιπόν ο κοινός μας στόχος, σύντομα να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική Ε, λύση όλων των θεμάτων που εκκρεμούν. Συμφωνία λοιπόν που θα μας επιτρέψει να περάσουμε και στη λύση των επόμενων θεμάτων που ακολουθούν όσον αφορά όλες αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιό παρακαλώ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εργάζομαι στην Γενική Διεύθυνση ε, Δικαιοσύνης. Σας ε, ευχαριστώ που μου δίδετε το λόγο για να μιλήσω για αυτό το θέμα. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής πρόκειται για μία, ε, ένα θέμα το οποίο χρονίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό και αφορά τα δικαιώματα ε, μετάφρασης και διερμηνίας. Ξέρουμε ότι καταρχάς το θέμα, με το θέμα της, ε, του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το οποίο είναι μία ε, επιτυχία στην Ευρώπη και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει διαδικαστικά να δοθούν κάποια ελάχιστα κοινά δικαιώματα σε όλους για να μπορέσουμε να έχουμε αγαστή συνεργασία, αναγνώριση όλων των αποφάσεων μεταξύ κρατών μελών και να προωθήσουμε την συνεργασία μεταξύ των ε, δικαστικών αρχών, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένης της μεγάλης κινητικότητας ε, των πολιτών μας ε, οι οποίοι ενδεχομένως στο εξωτερικό μπορεί να αντιμετωπίσουν μια τέτοιου είδους δικαστική διαδικασία. Τι θέλουμε πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε ε, δίκαια δίκη σε κάποιον ύποπτο ή κάποιον ο οποίος έχει συλληφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως θα θέλουμε να υπάρχει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Χάρτη Μελιωδών Δικαιωμάτων ο υψηλότερος δυνατός αριθμός, ε, βαθμός προστασίας των δικαιωμάτων όλων των εναγωμένων. Το 2009 αποφασίσαμε ότι τα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας θα πρέπει να τα και γι' αυτό το 2009 υποβάλαμε τον Ιούλιο την σχετική πρόφαση για την, πρόταση για την μετάφραση και την διερμηνία. Και μετά από την συνθήκη της Λισαβόνας, όπως ξέρετε, δεν εγκρίθηκε όπως ε, θα έπρεπε η, απόφαση δεδομένου ότι ε, δεν ίσχυε πλέον. Ο χάρτης πορείας, ο καινούριο καλούσε την Επιτροπή να νομοθετήσει για πέντε νέα θέματα όσον αφορά όλες τις διαδικασίες. Παρουσίασε λοιπόν μια νέα πρόταση η Επιτροπή για την ε, μετάφραση και τη διερμηνία βάσει της προηγούμενης πρότασης που κάνει και σύμφωνα με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά καθυστέρησαν τα πράγματα τότε γιατί δεν υπήρχε νέα επιτροπή. Τώρα σε χρόνο ρεκόρ μετά από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας επιτροπής και σύμφωνα με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας που άλλαξε κάπως τα πράγματα Κάναμε τη νέα πρόταση. Είπαμε ότι θα πρέπει ούτως ή άλλως οποιαδήποτε απόφαση να συνάδει με την νέα συνθήκη, με τα δικαιώματα σύμφωνα με την σύμβαση και βεβαίως χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα ε, ερμηνείας το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει κάποια κράτη-μέλη στο να πάρουν αποφάσεις που δεν θα είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων επίσης αποτελεί μέρος του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου και θα πρέπει όλες οι αποφάσεις να συνάδουν με τις σχετικές τους διατάξεις. Επίτροπος Ρέντινγκ είναι η νέα υπεύθυνη επίτροπος που ασχολείται με αυτά τα θέματα και παρουσίασε μία ε, πρόταση επιτροπή για να διασφαλίζεται ο, στο υψηλότερο βαθμό τα δικαιώματα των πολιτών καθώς και μετάφραση και σχεδιασμή και διάρκεια δικαστικών διαδικασιών. Είμαστε σίγουροι ότι η πρότασή μας ε, περνάει αν θέλετε τις εξετάσεις και στο Στρασβούργο, στο ε, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Σύμβαση. Θα πρέπει λοιπόν να πληρούνται κάποια κριτήρια και κάποιες απαιτήσει ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα κατάλληλα μέσα στη διάθεσή μας. Τρία σημεία στην πρόταση μας είναι πρωταρχική σημασίας και τα ανέφερε η Βαρονέσα Λότφορτ στην ε, παρέμβασή της, αλλά όπως ξέρουμε υπάρχουν και διαφορές. Το άρθρο 2 της πρότασής μας, το ε, δικαίωμα διερμηνής και μετάφρασης, χορηγείται στον ύπνο κατά τη διάρκεια των, ε, ε, των ε, συναντήσεων που έχει και ε, κατηδίαν με τον ε, δικηγόρο του πριν να έρθει η ημέρα της δίκης για να μπορέσει να προετοιμάσει αυτός πολύ καλά την υπράσπισή του. Επίσης, λέγουμε ότι η μετάφραση των κυρίων κειμένων θα πρέπει να παρέχεται γραπτός δηλαδή όλα τα σχετικά και σημαντικά έγγραφα της δικογραφίας, ώστε να μην επαφίονται όλοι μόνο σε μία προφορική μετάφραση της ε, τελευταίας στιγμής, δεδομένου ότι υπάρχουν στοιχεία και ματηρίες που πρέπει να υπάρχουν γραπτός στην ε, δικογραφία. Είναι κάπως διαφορετική άποψη εδώ της εισηγήτριας, δεδομένου ότι οι προτινόμενες τροπολογίες ε, δεν είναι και αντίθετο σε οποιοδήποτε συνοπτικά κείμενα. Στο άρθρο 3 επίσης λέγουμε ότι οποιοδήποτε ε, μπορέσει να ζητήσει απαλλαγή θα μπορεί να το κάνει έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί πλήρως για το τι σημαίνει αυτό. Όλα αυτά τα σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βεβαίω, η ποιότητα και η ουσία τη πρόταση μα ενδιαφέρει, συνεκτικότητα, σαφήνεια, φιλοδοξία, Αυτό είναι κάτι το οποίο μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η πρότασή μα λοιπόν είναι ε, χωρίς αμφισημίες, απολύτως σαφής και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών. Η πρόταση τη Επιτροπή αντικατοπρίζει ένα όραμα φιλόδοξο όλο αυτό το θέματο και πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται αυτή την άποψη, άρα χωρί έκπληξη βλέπουμε η πρόταση αυτή να αντικατοπνίζει το πνεύμα των τροπολογιών που κατέθεσε η εισηγήτρια Βαρονέ Σαλόντου. Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα είναι πρωταρχή σημασία και εμεί προσβλέπουμε σε συνεργασία ταχύτητα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που είναι οι συνομοθέτες ώστε να φτάσουμε σε ένα νομοθετικό κείμενο που θα εγγυηθεί όλα τα διαδικαστικά δικαιώματα ε, και την προστασία του υψηλότερου δυνατού επίπεδου έτσι όπως προβλέπεται στην, ε, στον χάρτη και την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βεβαίως με στενή συνεργασία και το Συμβούλιο θα εξετάσουμε όλα τα θέματα που έχετε θέσει. Θέλουμε να, προχωρήσει το θέμα σύντομα. Δεν θέλουμε να καθυστερήσει το πράγμα σε συνεργασία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και βεβαίως βασιζόμαστε στην εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι δύο προεδρήσεις, η Σουηδική και η Ισπανική, θέλουμε να καταλήξουμε σε ταχεία ε, υιοθέτηση της οδηγίας μετά από την πρώτη ανάγνωση τον Ιούνιο του 2010 και, ε, του 2010 και συμπληρωματικά θα πω ότι η Επιτροπή ήδη εργάζεται για το επόμενο μέτρο που προβλέπει στον οδικό χάρτη που είναι πρόταση για το δικαίωμα ενημέρωσης, το μέτρο Β όπως προβλέπετε που θα σας υποβληθεί το καλοκαίρι και ξέρουμε ότι η Επιτροπή σας ασχολείται με αυτά τα θέματα και μας προσθέτει για να υπάρχει η υψηλότερου δυνατού επίπεδου ε, προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Αντωνέσκου. Αρχίζουμε την συζήτηση. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Λάντφορτ είπε ήδη ότι βρισκόμαστε ενώπιον νέας κατάστασης. Υπάρχουν νέες διαδικασίες ε, που τίθενται σε ισχύ μετά την συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, τώρα έχει κατατεθεί η πρωτοβουλία, ασχοληθήκαμε με το έγγραφο και η έκθεση της κυρίας Λάντφορντ στηρίζεται στην πρωτοβουλία αυτή. Την περασμένη εβδομάδα κατετέθη η έκθεση της κυρίας Λάντφορντ και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ χαιρετίζω την πρόταση της Κομισιόν γιατί αναμφίβολα έτσι αναβαθμίζονται τα πρότυπά μας σε σχέση με αυτά που ίσχυαν στα πλαίσια της πρωτοβουλίας των κρατών μελών ε, επί της οποίας κινούμεθα μέχρι τώρα. Η κυρία Λάντφορντ και οι εκπρόσωπος της Κομισιόν το ανέφεραν αυτό. Μιλάμε για διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται για να καλυφθούν οι συνομιλίες δικηγόρου, υπόπτου, μετάφραση των σημαντικότερων εγγράφων. Γιατί η προφορική ε, σύνοψη δεν επαρκούσε. Μετά νομική ε, διαβούλευση, αν κάποιος θέλει να ε, παραιτηθεί από τα δικαιώματά του κλπ. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε το καλύτερο δυνατό κείμενο που θα ενισχύει τα δικονομικά δικαιώματα στις διαδικασίες και που θα ενισχύσει τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Ε, γι' αυτό χαιρετίζω το κείμενο της Κομισιόν, είναι πολύ καλύτερα τα πρότυπα. Ανησυχώ όμως για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι την έγκριση χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη, η γνωμοδότηση των Εθνικών Κοινοβουλίων και υπάρχει και η ρήτρα αυτοεξαίρεσης, opting out. Η Κομισιόν τι λέει για όλα αυτά. Νομίζω ότι μια ισορροπημένη προσέγγιση θα ήταν να ασχοληθούμε ταυτόχρονα και με τα δύο κείμενα, και με την έκθεση και με το κείμενο της Κομισιόν και με το κείμενο των κρατών μελών. Επίσης, το ψήφισμα για την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη αυτών των δικαιωμάτων, νομίζω ότι τα μέτρα που προβλέπει το ψήφισμα είναι πολύ σημαντικά και εδώ, γιατί αφορούν την ποιότητα. Πρόκειται για την αναγνώριση εμπειρογνωμόνων. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε και αυτό το θέμα υπόψη για να αποφανθεί το Κοινοβούλιο και από αυτού. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε θεσμικά να συμφωνήσουμε για να τα καταφέρουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκοέλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την Βαρόνι Λάτφορτ σε τρία σημεία και δεν συμφωνώ απόλυτα στο τέταρτο. Με το τέταρτο, συγγνώμη. Ποια είναι τα σημεία με τα οποία συμφωνώ και θα ήθελα να τι απαντήσω φόρο τιμή, διότι η θέση τη είναι πάρα πολύ συνεκτική και είναι πιστή σε αρχέ τι οποίε προσυπογράφουμε. Πρώτα απ' όλα, όταν λέει η Βαρόνι Λάντφορ ότι θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των πολιτών, θα πρέπει να είμαστε σαφεί. Πολλέ φορέ Μιλούμε για δικαιοσύνη, ελευθερία, δημοκρατία, αλλά πιο γρήγορα βρίσκουμε λύσεις ε, σε θέματα ασφάλειας παρά σε θέματα δικαιοσύνης, κοινέ λύσεις. Ό,τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών στον τομέα της δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να πω ότι είναι στην, ε, στην ε, πρώτη σειρά της μάχης υπέρ της περάσεων των δικαιωμάτων η Βαρόνη Λότφορντ όσον αφορά την ε, διάφορες ποινικέ διαδικασίες και τα δικαιώματα των πολιτών και τη διάρκεια της ποινική διαδικασίας. Το είπα πάρα πολλές φορές και το είπα στην τελευταία σύντηση που κάναμε στην Ολομέλεια ότι τα, οι ποινικέ διαδικασίες δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στο θέμα της μετάφρασης ή της διερμηνίας. Θέλω να έχουμε μία ευρύτερη έννοια και αντίληψη όσον αφορά τα δικαιώματα αυτά. Πότι πρώτη εδώ. Τρίτον, σημείο στο με το οποίο συμφωνώ. Η αξιολόγηση της θέσης των κρατών μελών. Λέει ότι είναι ανεπαρκής η πρόταση και εγώ συμφωνώ. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Η πρόταση της Κομισιόν είναι πολύ καλύτερη από την πρόταση που κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία σημεία με τα οποία συμφωνώ και τώρα θα σας πω που διαφέρουν οι απόψεις μας. Στην όλη διαδικασία. Υπάρχει μία σύγχυση που μας οδηγεί σε δύο πρωτοβουλίες. Μία και οι προτάσεις. Μία εκ μέρους της Επιτροπής, μία εκ μέρους των κρατών άλλων. Τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε μπορούμε να έχουμε και τα δύο αυτά προτάσει ε, μπροστά μα και να δουλέψουμε βάσει και των δύο. Ή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που συνήθω ακολουθούμε, να επιλέξουμε μία από αυτές. Θα, θα ήθελα λοιπόν εγώ να διευκρινίσουμε κάποια θέματα. Δεν θέλω να απορρίψουμε την πρωτοβουλία τη Κομισιόν. Θα ήταν λαθασμένο να την αγνοήσουμε για πολλού λόγου, αλλά κυρίω γιατί είναι καλύτερη από τι άλλε. Εάν έπρεπε εγώ να επιλέξω, θα προτιμούσα να δουλέψω με βάση την πρόταση της Επιτροπής. Για τρεις λόγους που θα σας εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, διότι δίνουμε ένα μήνυμα στους πολίτες μας. Εάν θέλουμε να έχουμε καλύτερες εγγυήσεις κατά τη διάρκεια της ποινική διαδικασίας θα πρέπει να βασιστούμε στην πρόταση που κατά την άποψή μου είναι καλύτερη για μας. Δεύτερον, για τις διαπραγματεύσεις. Όπως όλοι ξέρουμε και το ξέρει και η Βαρόνι Λάτφορτ, διότι έκανε εξ ονόματό μας πολλές και καλές διαπραγματεύσεις, είναι πιο εύκολο να διαπραγματευτεί κανείς με την Κομισιό και με το Συμβούλιο όταν η βάση εργασία είναι, ε, ε, προσεγγίζει περισσότερο αν θέλετε τις θέσεις μας. Και βεβαίω είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσουμε σε καλά αποτελέσματα όταν η βάση είναι πολύ, πολύ πιο μακριά από τι δικές μα θέσει. Στα πλαίσια λοιπόν της διαθεσμικής συνεργασίας θα πρέπει να είναι μαζί η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Τώρα, είναι διαφορετικές ε, οι νομοθεστικές της αρμοδιότητες της Κομισιόν, εάν πρόκειται για δική της πρωτοβουλία ή όχι. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να βρούμε μια λύση που θα υποτιμήσει την δυνατότητα παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην νομοθετική διαδικασία. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι για τους οποίους κύριε Πρόεδρε εγώ θα ήθελα να τονίσω περισσότερο την σημασία της πρωτοβουλίας που μας παρουσίασε η Κομισιό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουσούτιλ. Σάιμον. Σάιμον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Βαρόνι Λάντφορτ και να την διαβεβαιώσω ότι δεν είναι καθόλου ε, απλοϊκή η προσέγγιση της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την μακρά ενασχόλησή της με το θέμα. Συμφωνώ όμως με τους προηγούμενους δύο ομιλητές σχετικά με το τι δέον γενέστε. Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ το θέμα. Πρόκειται για ε, μια πρώτη περίπτωση μπορεί να επαναληφθεί. Έτσι εμείς ενδεχομένως θα δημιουργήσουμε προηγούμενο. Έχουμε δύο ανταγωνιζόμενες ε, προτάσεις και καλούμεθα να διαλέξουμε μία και να συνεχίσουμε με αυτήν. Καλό είναι αυτό, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι ποιο είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες μας εις ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους. Επί της ουσίας, νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν και όχι του Συμβουλίου είναι εκείνη η οποία προβάλλει ένα σαφές μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέξουμε πολύ πώς θα ε, χειριστούμε το θέμα, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον και κατά το χειρισμό του θέματος οι προτεραιότητές μας πρέπει να μπουν σε μια σειρά και νομίζω ότι το πρώτο μέλημα είναι η, ε, τα, δικαιώματα των πολιτών. Η Βαρόνι Λάντφορντ αυτό προσπάθησε να κάνει, να βάλει πρώτα τα δικαιώματα των πολιτών. Όμως ε, είναι σαφές, δεδομένων των συνθήκων, ότι η πρόταση της Κομισιόν δημιουργεί περισσότερη προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με την πρόταση του Συμβουλίου. Πιστεύω λοιπόν ότι θα αξίζει να δούμε επί της ουσίας την πρόταση της Κομισιόν. Άρα, ένα πράγμα μένει ακόμη. Πώς θα το κάνουμε διαδικαστικά. Δεν έχω σαφή απάντηση στο ερώτημα αυτό. Γνωρίζω όμως ότι είναι προτιμητέα η πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρομέρο Λόπε. Θα ήθελα και εγώ να σας πω την άποψή μου για την πρόταση της ε, Επιτροπής, για το κείμενο της Επιτροπής δηλαδή, που έχουμε μπροστά μας και θα ήθελα μετά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κόλιο και ο κύριος Μπουσούτη να προσθέσω το εξής. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε προτάσεις οδηγιών οι οποίες κάποια στιγμή σταμάτησαν δεδομένου ότι τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Θα έπρεπε η όλη διαδικασία να είχε ολοκληρωθεί, αλλά δεδομένου ότι τώρα ζούμε μια νέα κατάσταση, σταμάτησαν οι διαδικασίες. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε τώρα με μια εντελώς καινούρια κατάσταση και πιστεύω ότι με νέο τρόπο θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι οι θέσει των κρατών μελών, η πρόταση των κρατών μελών δεν σημαίνει ότι υποτιμούμε την πρόταση της Επιτροπής. Διότι και η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να συζητηθεί μαζί με τις προτάσεις των κρατών μελών δεν έχουμε να κάνουμε με μια συνήθη κατάσταση, με μια έκτακτη κατάσταση και θα πρέπει ε, ως έκτακτη κατάσταση να την χειριστούμε. Όπως είπε πάρα πολύ σωστά η εκπρόσωπος της Επιτροπής, έχουμε κάποιες εγγυήσει ε, κατά τη ε, διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, οι οποίες χρειάστηκε να τεθούν σε εφαρμογή μετά από την θέση σε ισχύ του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης έχουμε ένα κείμενο της Επιτροπής που βελτιώνουν τις εγγύησει Αλλά αν δεχθούμε το κείμενο τη Επιτροπής και αφήσουμε κατά μέρο την πρόταση των κρατών μελών, αναμφίβολα αυτό θα σημαίνει παράλυση του όλου θέματος, το οποίο είναι πήγον δεδομένου ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ισορροπία μεταξύ ε, των δικαιωμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης όπως και των δικαιωμάτων και των εγγύσεων που δίνουν στον τομέα της ε, ασφάλειας όπως είπε και ο κύριος Κουέλιο. Δίδονται κάποιες εγγύσεις από το πρώτο της Επιτροπής προβλέπονται βελτιώσεις και αλλαγές με τις τροπολογίες της ηγήτριας και με δικές μας τροπολογίες που θα πρέπει να μπορέσουν να κατατεθούν μέχρι το τε... τη λήξη της προθεμίας για να βελτιωθεί όλη η διαδικασία. Διότι όντως το 2004 η Επιτροπή επέβαλε την πρόταση αυτή, αλλά βεβαίως αυτή τη στιγμή η Πομισιό δεν θα έπρεπε να πει ότι στις προτάσεις της δεσμεύεται από τον ε, χάρτη πορείας. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε για να εξασφαλίσουμε όλα τα δικαιώματα και τις εγγύσεις που μπορούμε κατά τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών. Επιλέξαμε να συνεχίσουμε με το χάρτη πορείας. Έχουμε ένα πρώτο δικαίωμα, αλλά η κατάσταση αυτή έχει δημιουργηθεί από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι μια νέα κατάσταση, μια αρχική κατάσταση. Γι' αυτό θα ήθελα οι συνάδελφοι που έλαβαν το λόγο να το λάβουν αυτό υπόψη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με το κείμενο της Βαρόνης Λούτφορτ και να μπορέσουμε σύντομα να καταλήξουμε συμφωνία για το όλο κείμενο. Γιατί διαφορετικά θα παραλύσουμε όλη την διαδικασία και όλο το ε, πακέτο εγγυήσεων που παρουσιάζει η Κομισιόν και βελτιώνουν το κείμενο, τι θα γίνει. Ήδη συζητήσαμε αυτά τα τρία θέματα τα οποία παρουσιάζει ως βελτίωση πρότασή της Κομισιόν. Και στην πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει δεν ήταν απολύτως σαφής. Εγώ Χαιρετίζω το ότι διόρθωσε τη θέση της η και το, η πρότασή της βελτιώνεται. Αλλά βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση και πραγματικά εάν θέλουμε να προσπίσουμε τα δικαιώματα και διάρκεια των ποινικών διαδικασιών θα πρέπει η όλη διαδικασία να επιταχυνθεί και να μην αφήσουμε εντελώς κατά μέρος τις ε, προτάσεις που κάνουν τα κράτη-μέλη. Γιατί και παραλαμβάνω και πάλι θα παραλύσουμε την όλη διαδικασία. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω την πρωτοβουλία και των κρατών μελών και της Κομισιόν και πιστεύω ότι μπορούμε να, από τα δύο αυτά κείμενα να καταλήξουμε σε κάτι συμπληρωματικό. Ευχαριστώ. Κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι αυτονόητο και σωστό ότι ένα ύπνο και κατηγορούμενο πρέπει να έχει το δικαίωμα διερμηνία και μετάφραση όταν το χρειάζεται. Σε αυτό συμφωνώ με την πλειοψηφία των συναδέλφων. σω υπάρξει ανάγκη όταν ένα πρόσωπο μετακινείται από μία χώρα σε άλλη και εκεί υπόκειται στο νέο ποινικό σύστημα που είναι αναγκαίο, συχνά όμως είναι ένα από τα στοιχεία κόστη, μαζική μαζικής του που το παραβλέπουμε. Υπάρχουν όμω και άτομα που μετακινούνται λόγω σύλληψη, χωρίς να θέλουν δηλαδή. Βέβαια, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού του εντάλματο, γιατί υπονομεύει την εθνική επικυριαρχία και επιτρέπει έκδοση ατόμων για άτομα που δεν είναι ε, αδίκημα στη χώρα που τα εκδίδει. Ωστόσο, ακόμα και αν από λάθο γίνει, δεν θα ήταν προτιμότερο υποχρεωτική διερμηνία και μετάφραση να προηγηθεί τη σύλληψη και όχι να ακολουθήσει, αν ακολουθήσει. Ίσως η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να ισχύει και για περιπτώσεις ε, που δημιουργούνται από το Ευρωπαϊκό Έντερμα Σύλληψης και το κείμενο των κρατών μελών να ισχύσει για τις άλλες περιπτώσεις. Αυτό σας το δίνω σαν πρόταση να το σκεφτείτε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Σαρζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την συνάδελφο τη Σκιώδη των Πρασίνων που απουσιάζει, αλλά θα μιλήσω ξανά ονόματός της. Συγχαίρω και το σέβομαι στην κυρία Λάτφορντ για την πολύ σοβαρή δουλειά που έκανε. Είναι ένα θέμα που όντως αφορά την Επιτροπή μας. Μιλάμε για δικαιοσύνη, αλλά καλό θα είναι ο κόσμος να καταλαβαίνει για ποιο λόγο δικάζεται όταν δικάζεται. Γι' αυτό είμαστε υπέρ της μεθόδου και πρότασή σας. Ούτε θα αντιδικήσουμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν, γιατί τελικά το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να καταλήξει συμφωνία με το Συμβούλιο. Ταυτόχρονα έχει δίκιο η συγγήτρια που λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο της πρότασης της Κομισιόν. Η πρόταση αυτή είναι συνέχεια ενός ε, σχεδίου ε, πλαισίου απόφασης για ελάχιστες προδιαγραφές για τα δικαιώματα διαδικασίας από εργασία που είχε κάνει ο παλιότερο βουλευτής Μπέκινγκ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βάσο. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω επί της ουσίας, όχι επί της διαδικασίας. Μπορώ να μιλήσω τώρα. Θα ήθελα να εστιάσω στο πεδίο εφαρμογή. Ιδιαίτερα το άρθρο 1 παράγραφος 3 της ρυθμίσης που προτείνεται και να τονίσω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε ε, τις ποινικέ διαδικασίες από τις διαδικαστικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί τα περισσότερες διαδικασίες είναι ίσονος σημασίας ε, παράνομο παρκάρισμα, δεν είναι ποινικέ διαδικασίες. Γι' αυτό το άρθρο 1 παράγραφος 3 έχει μεγάλο νόημα, διότι η διερμηνία και η μετάφραση δεν μπορεί να διασφαλίζεται στη μεγάλη, ε, στο, μεγάλο αριθμό των ε, προσφυγών και διαδικασιών και επίσης ε, η απόφαση από 21 Δευτέρου του 84 του Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων είναι σημαντική. Δεν μπορούμε δηλαδή να ποινικοποιήσουμε σε αυτό το τομέα ε, ίσονο σημασίας διαδικασίας για να είναι πρακτική εφαρμογή του μέτρου από τα κράτη-μέλη, να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για όλους τους ενδιαφερομένους και να μην αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο που θα τον αντιμετωπίζαμε αλλιώ, να ε, μην μπορούμε να καλύψουμε όλες αυτές, όλο το μεγάλο αριθμό των διαδικασιών, διότι θα ε, έπρεπε να διπλασιαστούν τα πρόστιμα στην περίπτωση αυτή. Ε, ούτε ε, βεβαίως αυτό θα, ε, θα έβρισκε σύμφωνο τον Ευρωπαίο πολίτη τον διπλασιασμό μέσω, λόγω των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ προσεκτικά τα θέματα αυτά και να ξεχωρίσουμε από το μεγάλο αριθμό των διαδικασιών τις πραγματικά σημαντικές ποινικέ υποθέσεις και διαδικασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σταβάρης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως σκιώδης ήδη πήρα μέρος στους προηγούμενους τεμερείς διαλόγους πριν τη Λισαβόνα σχετικά με την έκθεση και γκρόσο συμφωνώ με την εισηγήτριά μας. Πολύ σωστά μερικά περίπλοκα προβλήματα ο ορισμός, γλωσσικά προβλήματα, πότε μια γλώσσα είναι μητρική γλώσσα ή πιο κατάλληλη γλώσσα προς μετάφραση. Πότε θα ζητήσει ή δεν θα ζητήσει το άτομο την ε, μετάφραση κλπ. Για το περιεχόμενο λοιπόν γενικά συμφωνώ με την προσέγγιση της συγκήτριας. Το πρόβλημα σχετικά με την επιλογή του κειμένου της Κομισιόν ή του Συμβουλίου για τις επόμενες φάσεις, όπως είπε και ο Κάρλος Κοέλιο στην αρχή, όντως το κείμενο της Κομισιόν φαίνεται πιο πλήρες. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα καθυστερούσε το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων. διότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουμε αποφάσεις που ήδη θα έχουμε περάσει. Θα είχαμε καθυστέρηση. Και επειδή ο χρόνος εδώ μετράει, γιατί όλοι δεν μιλάμε αφηρημένα, θέλουμε να είμαστε συγκεκριμένοι. Πρέπει να προχωρήσει γρήγορα το θέμα αυτό αν η συγγήτρια δεχτεί να βάλει στην έκθεσή της τις καλύτερες ιδέες του κειμένου της Κομισιόν αυτό θα ήταν το ιδεώδες. Έχω εμπιστοσύνη στο ανοιχτό της πνεύμα και ότι θα το κάνει αυτό. Συμφωνώ όμως και με τη γενική ανάλυση που λέει ότι το κείμενο της Κομισιόν και η Κομισιόν έχει νέες αρμοδιότητες με βάση τη νέα συνθήκη η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να είναι ο προτιμησιακός εταίρος μας. για να έχουμε πιο πλήρες πακέτο. Υποστηρίζει λοιπόν τη συγγετριά μας. Κύριε Παπα-Νικολάου, κύριε Παπα-Νικολάου, σας παρακαλώ, έχετε το λόγο να είστε σύντομος ευχαριστώ τη Βαρόνι Λάνφορντ για την πολύ καλή ε, εργασία που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ε, σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό, έχω καλυφθεί από την κυρία Αντωνέσκου και από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ε, όταν έχουμε και ένα νέο κείμενο από την Επιτροπή, αν μη τι άλλο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ε, βεβαίως όμως είναι μείζον για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να μην χάσουμε χρόνο και να προστατέψουμε ε, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, αλλά και άμεσα τα δικαιώματα εκείνων που καλούνται να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Επί τη ουσία, ένα μόνο προβληματισμό θα ήθελα να κάνω σε σχέση με τι νέε προτάσει που έχουμε. Συζητάμε για διερμηνία σε σχέση με, και με τι ιδιωτικέ συναντήσει του κατηγορουμένου με του δικηγόρου. Και επειδή είμαι και εγώ δικηγόρο, θα ήθελα να το θέσω και στην εισηγήτρια ω προβληματισμό. Δεν θα νιωθά πολύ άνετα κάθε φορά συναντήσεις που, που έχει ο δικηγόρος με τον κατηγορούμενο να υπάρχει ένα διαφορετικό πρόσωπο το οποίο θα διερμηνεύει. Και δεν ξέρω αν με αυτή την διαρκή εναλλαγή προσώπων, γιατί θα έχουμε υποθέτω ορισμό ενός διερμηνέα κάθε φορά από κάποιο κατάλογο, όποιος είναι, διαθέσιμο, ε, όποιος είναι διαθέσιμος, δεν ξέρω κάθε φορά αν θα μπορούσε αυτό να διασφαλιστεί στον βαθμό που θα θέλαμε ή αν θα έπρεπε να ε, βρούμε κάποια διαδικασία ούτως ώστε να είναι κάθε φορά ο ίδιος ο διερμηνέας ή εν πάση περιπτώσει να ορίζεται έστω από το δικηγόρο. Ε, ως προβληματισμό το θέτω και επιφυλάσσουμε βεβαίω και για τη συνέχεια της συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά τη συζήτηση α ξανακούσουμε την εισηγήτρια, την κυρία Λάτφορ, την οποία και παρακαλώ να κάνει μια πρόταση επί της διαδικασίας και για το χρονοδιάγραμμα επίσης. πρόταση για υποβολή τροπολογιών. για να καταλήξουμε σε ικανοποιητική συμφωνία προς το συμφέρον και ικανοποίηση όλων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, επί της ουσίας, επικροτώ την υποστήριξη εκ μέρους των συναδέλφων, γιατί συμφωνούμε με την Κομισιόν ότι το μέτρο αυτό πρέπει να ελεγχθεί και ως προς τη χάρτη και ως προς το Στρασβούργο. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε αυτό που λέμε τα τελευταία δέκα χρόνια από τότε που έχουμε το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης. Η άποψή μου είναι ότι χρειαζόμαστε το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης συν, συν, πλας, δηλαδή μέτρα που θα αυξάνουν την ποιότητα του δικαιώματων για δίκαιη δίκη του κατηγορούμενου και παρακολούθησα περιπτώσεις εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλλοντο που δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένοι με τα δικαιώματα που τους δόθηκαν. Αυτό το μέτρο θα έπρεπε να, το, θα έπρεπε να είχε εγκριθεί εδώ και καιρό. να επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Ταβάρες και νομίζω οι συνάδελφοι συμφωνούν. Θέλουμε να πάρουμε τις πιο καλές ιδέες από το κείμενο της Κομισιόν. Στην ουσία λοιπόν του αυτού που θέλουμε να πετύχουμε και συνάδελφοι να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στην ικανότητά μας να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Μερικοί από εμά έχουμε εμπειρία από αυτό. Έχουμε θετικό ιστορικό εμένουμε στις θέσεις μας. Και πετυχαίνουμε μια καλή συμφωνία. Εχτό έχουμε κάνει αυτό στο παρελθόν με το Συμβούλιο. Είναι θετικό το ότι η Προεδρία αναγνωρίζει το πλήρη ρόλο της Κομισιόν. Κανένας δεν πρόκειται να παρακάμψει την Κομισιόν ως προς το ρόλο της και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η πρόθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Πρόθεση λοιπόν του Συμβουλίου και δεν θα παίξουμε παιχνίδια εδώ. Αν και διαδικαστικά και θα επανέλθω σε αυτό, κινούμαστε με βάση το κείμενο των κρατών μελών, στην ουσία θα εμπνευστούμε, θα δανειστούμε ιδέες από την Κομισιόν και από απαλού και οι δικές μας τροπολογίες φυσικά και θα κάνουμε σκληρό παζάρι θα έχουν σκληρό αντίπαλό τους απέναντι το Συμβούλιο. Διαδικαστικά θα κινηθούμε με βάση το κείμενο του Συμβουλίου, αλλά δεν δεχόμαστε το κείμενο του Συμβουλίου, να γίνεται αυτή η διάκριση. Δεν δεχόμαστε το κείμενο της 23ης Οκτωβρίου 2009 για τη διαδικασία. Πρέπει να το συζητήσουμε κι άλλο με τους συναδέλφους. Απογοητεύτηκα λίγο για το ότι ζήτησα τη γνώμη των συναδέλφων για τη διαδικασία δεν είχα feedback από αυτούς που σήμερα διαφώνησαν. Αυτό δεν βοηθάει για πολύ βέβαια. Με απασχολεί το θέμα των, της περιπλοκής των καθυστερήσεων που μπορεί να δημιουργηθούν. Κείμενο της Κομισιόν σημαίνει ότι η περίοδο ε, μελέτης από τα Εθνικά Κοινοβόλια πρέπει να ξανανοίξει και αν θέλουμε να δουλέψουμε τυπικά με βάση το κείμενο της Κομισιόν η περίοδος για τα κράτη-μέλη που ε, ζήτησαν εξαίρεση θα πρέπει να ξαναρχίσει, να ξανανοίξει και δεν υπάρχει εγγύηση για το που θα καταλήξουμε γιατί όταν δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον να μελετήσει ένα θέμα μερικές φορές συμβαίνουν ατυχήματα γίνονται, παίρνονται διαφορετικές αποφάσεις Στις 8 Μαρτίου ο Υπουργός δικαιοσύνη Τζακ Στρό στο Ηνωμένο Βασίλειο υπόγραψε opt-in για το Ηνωμένο Βασίλειο επιέτη το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κατά της απόφασης πλαίσιο και τώρα έχουμε αυτή την απόφαση. Στροφή 180 μοιρών. Και δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί και άλλα εθνικά κοινοβούλια ξαφνικά να πούνε «Α, αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί και τώρα ας αλλάξουμε γνώμη». Δεν υπάρχει εγγύηση, καμία ότι θα συμφωνήσουμε τα μέτρα αυτά μέχρι τον Ιούνιο. Αν διαδικαστικά κινηθούμε με βάση το κείμενο της Κομισιόν. Επαναλαμβάνω όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραβλέπουμε το κείμενο της Κομισιόν. Θα μας είναι χρήσιμο να ενισχυθεί η ραχοκοκαλιά όλων και κοιτάω και προς το Συμβούλιο όταν το λέω αυτό Οι προφορικές συνόψεις, Φερρυπίν, oral summary. Μπορεί να πρέπει να το ξαναδούμε. Εγώ θα είχα διάθεση να συμβαστώ με το Συμβούλιο γι' αυτό. Με, αυστηρές, με αυστηρούς όρους βέβαια. Η, η κατεξαίρεση να επιτρέπεται. Μπορεί και η Κομισιόν έχει κάτι να μας πει γι' αυτό. Ο κύριος Μπουσουτήλ είπε μην τυχόν δημιουργήσει προηγούμενο αυτό. Όχι, όχι. Η κατάσταση είναι παράδοξη. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είναι ιδιόμορφη. Τέλος εντολής της ε, Κομισιόν, μεταβατική περίοδος. Δεν νομίζω ότι θα ξανασυμβεί αυτό. Και φυσιολογικά το Κοινοβούλιο προτιμάει πάντα την διαδικασία που στηρίζεται στο κείμενο της Κομισιόν ανέκαθεν. Ο κύριος Βός, ο κύριος Παπα-Νικολάου ανάφεραν ορισμένα σημεία. Θα ανταλάβω υπόψη τα σχόλιά σας. Χρειάζομαι να συζητήσω κι άλλο με τους συναδέλφους. Για να καταλήξω σε λύση που να τους ικανοποιεί όλους. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι το κείμενο της Κομισιόν δεν θα το παραμελήσουμε, δεν θα το παραβλέψουμε και θα το αναφέρουμε στο νομοθετικό μας ψήφισμα. Μεγάλο τμήμα του κειμένου της Κομισιόν με τον α το β τρόπο θα βρίσκεται στο τελικό κείμενο. Απλώς είναι μια τεχνικό διαδικαστικό θέμα. Από τη μια μεριά δεν είναι τόσο ζωτικό, από την άλλη μεριά είναι ζωτικό ως προς την επίπτωση που θα έχει στην, στις εθνικές αποφάσεις και στη διαβούλευση στα εθνικά κοινοβούλια. Και μακάρι να μην υπάρξουν επιπλοκές. Στο μεταξύ όλοι είμαστε ελεύθεροι να υποβάλουμε τροπολογίες και στο κείμενο της Κομισιόν. Ελπίζω με τις ε, συζητήσεις που θα επακολουθήσουν να είμαστε θέση για το επόμενο βήμα στις 7 Απριλίου αναγνωρίζοντας το ρόλο της Κομισιόν υπό την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ που προς μεγάλη ευγνωμοσύνη μας θα επιμείνει πολύ στο θέμα αυτό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι κάτι που εξάλλου θα περιμέναμε από την κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Λάντφορθ. Εκτιμούμε την πολύ λογική πρόταση που μας κάνετε. Ο συνήθως εξάλλου. Η συζήτηση ήταν αρκετά μακρά. Ακούσαμε τις διάφορες απόψεις. Η πρότασή σας είναι να το ξαναβάλουμε το σημείο στην ημερήσια διάταξη στις 7 Απριλίου συνεδρία στην Επιτροπή μας 7 Απριλίου για να έχουμε σύνθεση των θέσεων φυσικά και με την ενεργό συμμετοχή της ηγήτριας και των σκιωδών. Είδα ο πρόσωπος της Κομισιόν σήκωσε το χέρι για να μιλήσει. Επειδή όμως έχουμε καθυστερήσει, σας παρακαλώ συνεργαστείτε και μιλήστε την επόμενη φορά στις 7 Απριλίου αν συμφωνείτε. Δεν συμφωνείτε. Θέλετε να ξανανοίξετε το θέμα, Κομισιόν. Όχι, όχι, δεν θέλω να το ξανανοίξω. Ένα σύντομο σχόλιο. Δεν είναι θέμα επιλογής μεταξύ του κειμένου της Κομισιόν ή της πρωτοβουλίας των κρατών μελών. Δύσκολη κατάσταση και εκτιμώ το ρεαλισμό της Βαρονέσης Λάνφορ. Αν θέλουμε να εμπνευστούμε από την πρόταση της Κομισιόν, γίνεται, επειδή έχει γίνει σοβαρή δουλειά, να καταλήξουμε σε μία έκθεση που να καλύπτει και την πρόταση της Κομισιόν και την πρωτοβουλία των κρατών μελών. Μερικοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στα εθνικά κοινοβούλια. Εμείς ουσιαστικά υποβάλαμε μία λισαβονοποίηση μιας προηγούμενης πρότασης. Αν λοιπόν σε μία έκθεση δημιουργήσουμε συγχώνευση των δύο κειμένων θεσμικά θα είναι σωστή η λύση και δεν δημιουργείται και προηγούμενο για το μέλλον. Και δεν καθυστερούμε έτσι. Έχει οριστεί το χρονοδιάγραμμα και από το Κοινοβούλιο και από την Προεδρία και το τηρούμε. Απλώς χρειάζεται λίγη περισσότερη προετοιμασία με βάση τα δύο κείμενα. Πρόεδρος, δυστυχώς ξανανοίξατε τη συζήτηση. Παρακαλώ να μείνετε στο λογικό συμπέρασμα που πρότεινε η κυρία Λάντφορ. Η κυρία Λάντφορ ζήτησε το λόγο. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας. Να μην καθυστερούμε. Λάντφορ. Το δικό μου συμπέρασμα και της Κομισιόν δεν είναι το ίδιο και νομίζω η Επιτροπή μας συμφώνησε με τη δική, μας, με τη δική μου πρόταση και όχι με της Κομισιόν. Με όλο το σεβασμό που τις έχω. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο η Κομισιόν. Δεν θα συγχωνεύσουμε τα δύο κείμενα. Εγώ είπα, τυπικά διαδικαστά θα κινηθούμε βάσει το κείμενο των κρατών μελών, αλλά θα εμπνευστούμε από το κείμενο της Κομισιόν όσον αφορά την ουσία. Είναι δύο διαφορετικές μέθοδοι αυτές και έχω σοβαρούς διαδικαστικούς λόγους να προτείνω αυτό που πρότεινα. γιατί επιπλοκές και καθυστερήσεις από τη συγχώνευση των δύο κειμένων καταρχήν δεν ξέρω αν γίνεται σε μια έκθεση αυτό θα δημιουργήσει επιπλοκές στις εθνικές πρωτεύουσες σε μερικές εθνικές πρωτεύουσες άρα αυτό που είπε η Κομισιόν δεν μας βοήθησε και πολύ να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και παρακαλώ την Κομισιόν να συμφωνήσει με το δικό μου πόρισμα Πρόεδρος, μάλιστα ακούσαμε την πρότασή σας, έγινε δεκτή από την Επιτροπή ΛΙΜΠΕ. Συμφωνούμε λοιπόν να μπει το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη στην επόμενη συνάντησή μας 7 Απριλίου. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο. Προχωρούμε τώρα στο σημείο 13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 Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Παρακαλώ λοιπόν, ε, εάν παραμείνετε στην αίθουσα, να υπάρχει ησυχία. Παρακαλώ πολύ. Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι εδώ ακολουθούμε την προθεσμία που έθεσε ο πρόεδρος κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕΣ στις 4 Μαρτίου για να ενημερωθεί εάν τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ επιθυμούν να αντιταχθούν στο μέτρο. Οι συντονιστές τεσσάρων πολιτικών ομάδων, ΕΛΚ, ε, Φιλελεύθεροι, ε, συντηρητικοί μεταρρυθμιστέ και πράσινοι απάντησαν εξ ονόματο των ομάδων ότι θέλουν να αντιταχθούν στο μέτρο. Ο εισηγητή, ο κ. Μάικλ Κάσμαν, ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση της 4 η Μαρτίου ότι η σύστασή του είναι όχι αντίθεση στο μέτρο που σχεδιάζεται. Προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε ως εξής. Πρώτον, θα ερωτήσω τα μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ αν στηρίζουν ή όχι την πρόταση του εισηγητή. Δεύτερον, αν η σύσταση του εισηγητή δεν γίνει δεκτή, θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία επί σχεδίου ψηφίσματος με το οποίο η Επιτροπή μας θα συστήσει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αντιταχθεί στο σχεδιαζόμενο μέτρο εξηγώντας τα, τους βασικούς λόγους της αντίθεσης το κείμενο που έχει διανεμηθεί κατετέθη από τη Γραμματεία λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες συζητήσεις. Σημειώστε παρακαλώ ότι το ψήφισμα θα πρέπει να σταλεί στην Ολομέλεια ε, της 24 η 25 η μαρτιου 2010 ώστε να εγκριθεί πριν λήξει η προθεσμία του Κοινοβουλίου στις 7 Απριλίου 2010. Κύριε Κάσμαν, ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προχωρήσουμε με ησυχία γιατί αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως και πολλά άλλα της Επιτροπής μας. Θέλω λοιπόν η, ε, το συμπέρασμα να στηρίζεται σε στοιχεία. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται σε δύσκολη θέση και δεν μας βοήθησε η διετή συζήτηση του Συμβουλίου, η οποία επίσης ήταν δυσχερής και προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα αυτό. Η νομική γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου Ευχαριστώ. Ε, την οποία σέβομαι ιδιαίτερα είναι ότι τα μέτρα ξεπερνούν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12.5 του κώδικα Σέγγεν επειδή δεν συνιστούν πρόσθετα μέτρα σχετικά με την επιτήρηση γενικότερα. Αυτό είναι μια πολύ ε, μικρή σύνοψη. Άρα λοιπόν η νομική υπηρεσία λέει να μην γίνει δεκτό γιατί ξεπερνά τις εξουσίες. Η Σεσίλια Μάλστρομ απέστειλε επιστολή επίσης εκφράζοντας διαφορετική γνώμη άρα έχουμε δύο διαφορετικές νομικές απόψεις, γνωμοδοτήσεις. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με την απόφαση και γι' αυτό θέλω να εγκρίνομαι την απόφαση, δηλαδή να μην εκφράσουμε αντίθεση στο μέτρο, το νόημα λοιπόν είναι να υπάρχει κάποια βεβαιότητα στις, ε, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σε σχέση όχι μόνο με την επιτήρηση αλλά και την ανάσχεση και διάσωση και αναζήτηση. Τώρα, να ξεκαθαρίσω τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να επαναληφθεί το περσινό δυσάρεστο θέαμα όπου δύο κράτη-μέλη αρνήθηκαν τη διάσωση ε, ανθρώπων από την Νότια Μεσόγειο γιατί δεν ήθελαν να ασχοληθούν με τα ανακύπτοντα προβλήματα της παράνομης μετανάστευσης ε, ή της πιθανής αίτησης ασύλου. Η της πιθανης σύμβαση ασυλου λοιπόν τι κάνει εδώ. Ε, φέρνει τη Διεθνή Σύμβαση στα πλαίσια του κοινοτικού κεκτημένου και διασφαλίζει έτσι τη συμμόρφωση και τον σεβασμό των διατάξεων ε, μέσω του ΔΕΚ. Είναι δύσκολη η θέση μας ε, γιατί τα μέτρα αυτά το Κοινοβούλιο τα ζητούσε και η κυρία Πλάσσερτε τα ξαναζήτησε στην ε, Επιτροπή αυτή του Κοινοβουλίου τελευταία φορά τον Ιανουάριο φέτος. Εν πολλής συνιστούν το, στο δεύτερο μέρος ε, τις υποχρεώσεις που πρέπει να σέβονται τα κράτη-μέλη βάσει διεθνών συμβάσεων και του δικαίου της θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή τη στιγμή δεν ε, εφαρμόζονται από το ΔΕΚ. Όταν όμως γίνει δεκτή απόφαση, τότε θα ε, είναι υπεύθυνο το ΔΕΚ. Η νομική υποχρέωση λοιπόν... Ε, έρευνας και διάσωσης, αν υπάρχει ανάγκη, αυτό γίνεται κάτι που δεν μπορεί να ε, αρνηθεί πλέον το κράτος μέλος. Όμως, το ηθικό δίλημα θα πούμε στο Συμβούλιο και την Κομισιόν είναι λάθος η νομική βάση, πάρτε την από εδώ. Νομίζω ναι. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα έρθει νέα πρόταση από την Κομισιόν. Είναι νέα η Κομισιόν, θα πρέπει πρώτα να συζητήσει τους κόλπους της και να καταλήξει σε νέα πρόταση. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα έρθει νέα πρόταση συμπεφωνημένη με το Συμβούλιο ε, ή το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της θητείας μας ε, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μπορεί πάλι να ανακύψουν φέτος το καλοκαίρι. Γι' αυτό λοιπόν, λόγω των εξαιρετικών αυτών συνθήκων και χωρίς να δημιουργείται κανένα προηγούμενο, γιατί θυμηθείτε ότι το προηγούμενο τίθεται μόνο αν το Κοινοβούλιο δεχτεί ότι αυτό που κάνει από είναι προηγούμενο. Αυτό ας το κρατήσουμε από τη μια. Και βεβαίως αν συμφωνήσουμε μπορούμε να εξειδικεύσουμε τη σύμφωνη γνώμη σας. Και γιατί πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν και με τρόπο κατεπήγοντα να προτείνουν μέτρα στα πλαίσια πρότασης ε, νομοθετικού περιεχομένου ή στα πλαίσια της αναθεώρησης του κώδικα του Σέγγεν ή στα πλαίσια του Frontex. Επίσης, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κρατήσει ανοιχτές όλες τις νομικές επιλογές που μπορεί να καταστούν αναγκαίες. Για να παραφράσω τη Βαρόνη Λάντφορντ, ε, αυτό ε, σαν μια προφορική σύνοψη. Συγγνώμη που μακρυμγόρησα, το συζητήσαμε αυτό στην πολιτική μου ομάδα και είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Νομίζω ότι έχω την υποστήριξη της πολιτικής μου ομάδας και καταλήξαμε εδώ μετά από σκληρό προβληματισμό ε, και αντιπαραθέσεις. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια πολιτική απόφαση για να λύσουμε το ηθικό αυτό δίλημα. Υπάρχουν μερικοί και νομίζω ότι θα πρέπει να το πω, υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι το μέτρο της ανάσχεσης ή αναχέτησης θα εμποδίσει από ορισμένους την ε, δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο. Εγώ δεν νομίζω ότι το μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά ε, ορισμένοι έχουν κάποιες τέτοιες ανησυχίες. Τελειώνω λοιπόν στο σημείο αυτό. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να επανέλθω με ερωτήσεις ε, και το αφήνω το θέμα στη σοφία της Επιτροπής αναγνωρίζοντας απόλυτα κύριε Πρόεδρε ότι όλες οι γνωμοδοτήσεις που ακούγονται εδώ και εκφράζονται εδώ και που θα εκφραστούν μέσα από την ψηφοφορία σήμερα έχουν την ίδια εγκυρότητα ε, και την ίδια υποστήριξη ε, εννοώ από αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε σύντομα την Προεδρία και την Κομισιόν. Ο κύριος Μπούργος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τρίτη φορά που στην Επιτροπή σας μιλούμε για αυτή την πρόταση απόφαση του Συμβουλίου που σας υπευλήθη εδώ και ένα χρόνο σχεδόν. Πιστεύω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το φάκελο. Από όσον βλέπω θα πρέπει να σας εξηγήσω γιατί υιοθήσαμε αυτή την πρόταση με αυτή τη νομική βάση. Διότι κατά τη δική μας άποψη ο, για τα σύνορα και τον κώδικα υπάρχουν διαφορετικά μέτρα που αφορούν την επιτήρηση των συνόρων που συμπεριλαμβάνουν στο άρθρο 18 και αφορούν την επιτήρηση μεταξύ συνόρων σε ανοιχτή θάλασσα συγκεκριμένη περίπτωση καθώς και, τα μέτρα που αφορούν τις επιθεωρήσεις που γίνονται στα σύνορα τα ίδια. Έχουμε διαφορετικά θέματα, διαφορετικούς στόχους και στον κώδικα ορίζονται διαφορετικά γιατί οι επιπτώσει τους είναι διαφορετικές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο κώδικας εγκρίθηκε μετά από τη διαδικασία συναπόφασης του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, γιατί ήδη ίσχυε τότε αυτή η διαδικασία. Και δεδομένου ότι πρόκειται για διαφορετικά μέτρα, το άρθρο 12 θεσπίζει κάποιες αρχές και λέει ότι μπορούν κάποια συμπληρωματικά μέτρα σύμφωνα με την διαδικασία της επιτροπολογίας να εγκριθούν. Αυτό είναι αυτό το οποίο πρότεινε η Επιτροπή και αυτό είναι βασικά ε, αυτό το οποίο έκανε με την υιοθέτηση κάποιων αλλαγών το Συμβούλιο. Κατά την άποψή μας αυτή λοιπόν είναι η σωστή νομική βάση και την αιτιολόγηση. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κατά την άποψή μας το θέμα που συζητείτε τώρα από τεχνικής απόψεως είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Γι' αυτό Υπήρξαν ε, εκτενέστατε συζητήσει μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή, καθώς και στην Επιτροπή που ασχολείται με τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας κόστησε πάρα πολύ να φτάσουμε συμφωνία, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι γιατί είναι πρώτη φορά που τέτοιου είδου θέματα διευθετούνται σε κοινοτικό επίπεδο. επίση θα ήθελα να τονίσω ότι αν τώρα δημιουργείται πρόβλημα κατά τη διάρκεια μίας ε, επιχείρησης θαλάσσιας με την Frontex δεν συμβαίνει και κάτι το σημαντικό. Δεν συμβαίνει τίποτε δεδομένου ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κοινοτικό δίκαιο που Εάν εγκριθεί η απόφαση θα υπάρχει ένα κοινοτικό πλαίσιο. Θα υπάρχουν επιπτώσεις που σε περίπτωση προβλήματος μπορούν να οδηγήσουν ανάλογα με το πρόβλημα ή σε ε, διαδικασία της κατά της Κομισιό ή σε μια διαδικασία ε, πιο στενού ελέγχου εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Ο υπεύθυνο ε, της πολιτικής ε, σύνορα μπορεί να κληθεί από σας και από το Συμβούλιο και να του ζητήσετε το λόγο. Γιατί ε, εφαρμόστηκαν οι κοινοτικοί κανόνες, ήταν οι σωστοί, γιατί καταλήξαμε σε αυτήν την απόφαση ε, να ζητήσετε κάποια αλλαγή. Προς το παρόν όμως πρέπει να πω ότι δεν εφαρμόζεται εδώ το κοινοτικό δίκαιο. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή έχει μία προστιθέμενη αξία και, και συνεισφέρει και στον δημοκρατικό έλεγχο που μπορεί να γίνει σε επίπεδο Frontex. Κατά την άποψή μου θα υπήρχε διακριτική ενταχείριση μεταξύ των ε, κοινοτικών οργάνων δεν υπάρξει συμφωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι κάτι που είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να δραματοποιούμε την κατάσταση, λοιπόν, επαναλαμβάνω, αν δεν υπάρχει συμφωνία προ το παρόν. Πιστεύω ότι θα επιληθούν τα προβλήματα. Από πρακτική πλευρά, η συνενετική λύση, αν χρειαστεί να καταλήξουμε σε αυτή, ούτε θα είναι σύντομη, ούτε εύκολη. Γιατί θα είναι σύντομη, διότι η όλη διαδικασία η εσωτερική κάθε θεσμικού οργάνου πρέπει να γίνει σεβαστή από τους άλλους και εσείς η και το Συμβούλιο και η Κομισιό και χρειάζεται αν φτάσουμε σε συμφωνία χρόνο για να το θέσουμε σε εφαρμογή. Βεβαίως δεν είναι εύκολο να υπάρξει και συμφωνία λέγω και βεβαίως δεν αναφέρουμε το τούτο στην Κομισιό ούτε σε εσά. Στο Συμβούλιο δεν υπήρξε ομοφωνία για την υιοθέτηση αυτής της απόφασης. Τώρα, εάν τεθεί εκ νέου το θέμα στους υπουργούς, θα ξανανοίξει η συζήτηση και η Κομισιό θα παρουσιάσει ή την ίδια πρόταση που έχει κάνει μέχρι τώρα ή κάτι διαφορετικό. Και το πιο πιθανό είναι ότι θα το συζητήσουν το όλο θέμα εκ νέου οι υπουργοί και λογικά θα υπάρξει μια κάποια διαδικασία επειδή δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Σα λέγω και πάλι δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Τελικά πιστεύουμε ότι η απόφαση είναι χρήσιμη και συνιστούμε να υιοθετηθεί. Βεβαίω, εδώ δεν προτείνουμε μια απόφαση που θα μας δώσει τη θαυματουργή λύση. Δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Πρώτη φορά για αυτό το θέμα προτείνεται κάτι το κοινοτικό. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι το χρήσιμο που θα βοηθήσει το σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα. Επίση, πρέπει να υπογραμμίσω ότι έχουμε πάρει πάρα πολλέ προφυλάξει. Είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα ήθελα να σα παραπέμψω σε διακήρυξη του Συμβουλίου όπου γίνεται λόγος για τον τρόπο τον οποίο εφαρμόζεται αυτή η, απόφαση και δίδονται και διάφορες Ενημερωτικέ εξηγήσει. Σα είπα, έχουμε προσέξει πάρα πολύ τα πράγματα σε αυτό το τομέα και όταν έρθει εδώ υπεύθυνο τη ε, Frontex, εσά ή σε κάποιο όργανο, μπορείτε να του κάνετε σχετικές ερωτήσεις. Τι είδου μέτρα πρέπει να λαμβάνονται από τώρα. Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για την θαυματουργή λύση όλων των προβλημάτων, αλλά πιστεύουμε ότι οι ε, θαλάσσιες, ε, επιτήρηση των θαλασσίων εξωτερικών συνέρων στο ε, Frontex θα γίνονται με καλύτερο δυνατό τρόπο με την εθέτηση αυτής της αποφάσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ακούσουμε την Επιτροπή να ακούσω και την άποψη των μελών, δεδομένου ότι θα πρέπει να ψηφιστεί το θέμα. Θα ήθελα, επειδή θα ψηφίσουμε, να ρωτήσω αν έχετε την ε, κάρτα σας για να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία ή διανατάσσεω χειρός να ψηφίσουμε. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βάσει της επιστολής της Επιτρόπου Μάλμστρομ στην Επιτροπή θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, σχετικά με τη νομική πτυχή. Η Κομισιόν είναι πεπισμένη ότι η νομική βάση και το προτινόμενο μέτρο είναι σωστά. Για την ιστορία, το Συμβούλιο επίσης συζήτησε μακρόν νομικά θέματα, αλλά με διαφορετικές ενστάσεις. Κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο ισχυρίστηκαν ότι δεν υπάρχει ε, ενωσιακή αρμοδιότητα σε αυτό το τομέα. Δεν υπάρχει ε, αρμοδιότητα της Ένωσης σε ό,τι αφορά έρευνα και διάσωση ε, μεταναστών που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Από την πλευρά της Κομισιόν θα πρέπει να πω ότι θεωρούμε κάπως λυπηρό το γεγονός ότι καθ' όλες τις συζητήσεις ε, επικεντρωθήκαμε σε νομικά θέματα και όχι σε πολιτικά. Δηλαδή την ανάγκη η Ένωση να φροντίσει ώστε να υπάρχουν κανόνες όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ε, απαιτητικό αυτό θέμα της μετανάστευσης στα εξωτερικά μας σύνορα. Επίσης με κάθε σεβασμό θυμίζω ότι το μόνο αρμόδιο θεσμικό όργανο για να λύνει τέτοιου είδους θέματα νομικά είναι το ΔΕΚ που σε τελευταία ανάλυση είναι το μόνο που μπορεί να πει, να αποφανθεί αν πρόκειται για τη σωστή νομική βάση ή όχι. Επί της ουσίας, ο εισηγητής ήδη έδωσε καλό παράδειγμα με ε, την έρευνα και τη διάσωση. Να δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα. Το θέμα της αρχής της μη επαναπροώθησης και η εφαρμογή της στα διεθνή ύδατα. Διευκρινίζω, από την πλευρά της Κομισιόν θεωρούμε ότι με βάση τον κώδικα του Σέγγεν, με βάση τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτή η αρχή εφαρμόζεται στην ανοιχτή θάλασσα. Όμως αυτή είναι μια ερμηνεία που αμφισβητείται και υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη, πολλοί οργανισμοί που θεωρούν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η απόφαση αυτή που διακυβεύεται σήμερα ε, ρυθμίζει άπαξ και διαπαντός αυτή την αμφισημία, διευκρινίζοντας ότι η αρχή εφαρμόζεται και μάλιστα δίνει οδηγίες σχετικά με το πώς θα εφαρμόζεται η αρχή αυτή στην πράξη. Τρίτον, για τον κανονισμό του Frontex. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν υπέβαλε πριν από δύο εβδομάδες μια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση, όπου κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν, βάλαμε εκεί ό,τι μπορούσαμε για να ενισχύσουμε την πτυχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τον οργανισμό Frontex. Ο κανονισμός όμως της Frontex ασχολείται με τη λειτουργία της υπηρεσίας και τις ε, αρμοδιότητές της. Ε, αυτή εδώ η απόφαση αφορά τις υποχρεώσει των κρατών μελών που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο και το διεθνέ δίκαιο. Και ερμηνεύει και διευκρινίζει πω αυτές οι ε, υποχρεώσεις θα τηρούνται στην πράξη. Οι δύο μηχανισμοί είναι συμπληρωματικοί και αμοιβαία απαραίτητοι. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή σχετικά με τις επιχειρήσεις του 2010. Από την πλευρά της Κομισιόν ανησυχούμε ιδιαίτερα. Θέλουμε οι επιχειρήσεις που έχουν σχεδιαστεί από τον Frontex στα νότια σύνορα να λάβουν χώρα, να πραγματοποιηθούν. Και σε ό,τι αφορά την προστασία των προσώπων, γιατί περί αυτού πρόκειται σε τελευταία ανάλυση, προστασία των δικαιωμάτων των ε, μεταναστών που κάτω από τραγικές συνθήκες προσπαθούν να προσεγγίσουν την Ευρώπη και την προθυμία των κρατών μελών να δεχθούν να συμμετέχουν στις ε, επιχειρήσεις του Frontex το 2010. Πολλά κράτη-μέλη είπαν δικαίως νομίζω ότι θα πρέπει μια τέτοια απόφαση να είναι προϋπόθεση για να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις του Frontex. Η απουσία της αποφάσεως δεν μειώνεται μόνο η, η δυνατότητα που έχουμε να προστατεύουμε ατομικά δικαιώματα, αλλά υποβαθμίζομαι και την ικανότητα της Ένωσης να αντιδρά στη μετανάστευση διαθαλάσσης και να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι εξ ονόματος του Επιτρόπου μου πρέπει να πω ότι το σενάριο συνεχιζόμενης απουσίας αυτών των κανόνων δεν θεωρείται ότι είναι πολιτική ε, ευθύνη της Κομισιόν και καλό την Επιτροπή να μην απορρίψει το σχέδιο απόφασης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστώ. Και τώρα αρχίζουμε τη συζήτηση. Ζανίν Χανής Πλάσερτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί μιλούν για τις ε, επιχειρήσεις του 2010 και την ευθύνη που έχουμε σε αυτά τα πλαίσια. Πραγματικά είναι τρομερό διότι είχαμε επιχειρήσεις κατά το παρελθόν όπου ε, τα κράτη-μέλη ε, δεν είχαν πρόβλημα να συνεχίσουν. Δεν πρέπει να ε, φορτίζουμε συναισθηματικά το θέμα λοιπόν. Χρειάζονται, συμφωνώ με τον εισηγητή, οι κατευθυντήριε γραμμέ, αλλά δεν έχουμε και μια αίσθηση τη πραγματικότητα. Όταν μιλάμε για αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και την ισχύ τους, δεν είναι δεσμευτικές. Οπότε το θέμα της λογοδοσίας των κρατών μελών πρέπει να εξεταστεί αφού δεν είναι δεσμευτικές οι κατευθυντηρίες. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των κατευθυντηρίων γραμμών, συμφωνώ ότι χρειάζονται, ε, ήδη το είπαμε αυτό, αλλά αμφισβητώ την ισχύ που έχουν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί με μεγάλη προσοχή. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε μια ξεκάθαρη γνωμοδότηση των νομικών υπηρεσιών επί του θέματος. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια νομική υπηρεσία έχει δίκιο. Να το δούμε ρεαλιστικά. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να συνδυάσουμε τις νομικές υπηρεσίες Κοινοβουλίου Κομισιόν, νομίζω ότι ε, υπάρχει επίσημη θέση του Συμβουλίου. Έχω συζητήσει με κάποια κράτη-μέλη και θεωρούν ότι η νομική γνωμοδότηση θα πρέπει να ενσωματωθεί, στο, δηλαδή να προσαρτηθεί στον κανονισμό ε, για τον Frontex. Πώς μπορεί να γίνει όμως αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχω. Αν συμφωνήσουμε δηλαδή τώρα, μετά τι θα γίνει. Η πολιτική μου ομάδα δεν θα εγκρίνει την πρόταση. Κάναμε μια έντονη συζήτηση στην ομάδα μου για να προετοιμάσουμε την ε, θέση μας κατά τη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Είναι δύσκολο θέμα, ιδιαίτερα, όπως ε, είπα, όταν κάποιος παίζει ε, το συναισθηματικό χαρτί. Δεν νομίζω ότι αυτό εξυπηρετεί το Συμβούλιο, να παίξει δηλαδή το χαρτί της συναισθηματικής φόρτισης στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ, κύριε Ρωμέβα. Ευχαριστώ πολύ. Κατανοώ απόλυτα τους λόγους και συμμερίζομαι τις ανησυχίες για τα ηθικά θέματα τα οποία ανέφερε ο συνάδελφος. Κάσμαν. Πρόκειται για δύσκολη απόφαση. Αυτό είναι θέμα το οποίο το συζητήσαμε και στη δική μου ομάδα και όντω πρόκειται για μία απόφαση που μας φέρνει αντιμέτωπους με πολιτική ηθική και νομική υφή θέμα. Είναι όμως απαραίτητο, κατά την άποψή μας, να έχουμε ε, συνεκτικότητα, αν θέλετε, σε αυτό το θέμα με τη θέση που έχουμε εκφράσει και για άλλα παρεμφερή θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η νομική βάση και που είναι η βάση της έκθεσης αυτής. Δηλαδή, εάν σε κάποια σημαντικά θέματα η έκθεση της νομικής υπηρεσίας και η απόφαση είναι σημαντική, θα πρέπει να την ακολουθήσουμε, διαφορετικά θα αποδυναμωθεί η θέση μας όταν συζητούμε παρεμφερή θέματα άλλες φορές. Όπως λέει και ο κύριος Κάσμαν, το ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε προηγούμενο δεν έχει καμία αξία, διότι ούτως ή άλλως θα δημιουργηθεί προηγούμενο. Η έννοια λοιπόν αυτή είναι κάτι το οποίο εν υπάρχει παρά το γεγονό ότι θέλουμε ή θα θέλαμε ή θα πούμε ότι δεν θα δημιουργήσει κάτι τέτοιο προηγούμενο. Άρα διαφωνώ και με την Κομισιό. Η διαδικασία είναι πολιτική. Δεν κάνουμε κάτι κατά της νομικής βάσης, απλώς πρόκειται για κάτι το οποίο είναι από άποψη πολιτικής πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη όμως, και ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να αναφέρω και το ανέφερε και η Ζανίν είναι το θέμα του δεσμευτικού χαρακτήρα αυτού της απόφασης. Θα είχαμε κάποια άλλη συζήτηση εάν δεν ήταν δεσμευτικό το άλλο θέμα. Άρα το ερώτημα το οποίο θέτουμε τουλάχιστον στην ομάδα είμαστε τι πραγματικά, πραγματικά θα αλλάξει στην πράξη, στην πρακτική, στην συγκεκριμένη δράση που αναλαμβάνεται συγκεκριμένα ζώνες η έγκριση αυτής της απόφασης δεδομένου ότι βασικά τα πάντα εξαρτώνται από την πολιτική βούληση των κρατών που θα υιοθετήσουν την απόφαση. Και όπως είπαμε, εδώ η βούληση τους εξαρτάται και από τις διεθνείς συμβάσεις που υπάρχουν. Άρα έχουμε αμφιβολίες για το εάν τώρα με την υιοθέτηση αυτής της απόφασης θα αλλάξουν πρακτικές οι οποίες είτε δεν πληρούνται είτε δεν υπάρχει βούληση, ε, ε, πολιτική βούληση να εφαρμοστούν. Η συζήτηση για τον ε, κανονισμό της Φρονκτέτ και του Θάλασσα νομίζω ότι μας δίνει τη δυνατότητα να ενεργήσουμε σωστά και να κάνουμε σωστά τα πράγματα. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι με απασχολεί κάποιος εκβιασμός ε, που γίνεται εθελούσια ή όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας λένε κάποιοι αν δεν ψηφίσετε το μπλοκάρετε. Αν ψηφίσετε άλλο διαφορετικό. Ακούω αυτά τα πράγματα για το θέμα αυτό εδώ και από το 2006 και μετά. Όλο αυτό τον καιρό δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα για να μπορέσουμε να θεσπίσουμε το σύνολο μέτρων που θέλουμε να θεσπίσουμε. Διότι κάθε φορά που πρέπει να τρέξουμε και να κάνουμε κάτι, μας ε, την τελευταία στιγμή η ευθύνη πέφτει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω όμως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι θα ενεργήσουμε σωστά και να μην μας γίνεται ηθικός εκβιασμός κατά κάποιο τρόπο. Το περιεχόμενο δεν μας ενθουσιάζει, αλλά πρέπει να πω ότι από θέμα ε, από την οπτική γωνία της ευθύνης εμείς αποφασίσαμε να απορρίψουμε αυτή την πρόταση που γίνεται από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Σας απειλώ λέει ο κύριος Ντία Πρέπει να λάβω θέση και να εξηγήσω τη θέση μου διότι όπως ξέρουν κάποιοι από εσά, το θέμα αυτό που αφορά τη Frontex είναι ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Θα ψηφίσω όπως η ομάδα μου και με απόλυτη σαφήνεια πρέπει να σας πω ότι είμαι υπέρ της, ε, της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για ποιο λόγο τη διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά το άρθρο 12 του κώδικα των συνόρων και τα πέντε του σημεία δια, μελέτησα πάρα πολύ προσεκτικά τις παρατηρήσεις της Επιτρόπου Μάλστρομ και επαναλαμβάνω την έκθεση νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να πιστεύω την προσοχή στα εξή θέματα. Πρώτα απ' όλα, σε αυτή τη συζήτηση, στο σημείο 4 του 12 του κώδικα και στο σημείο 5 που δίνει κάλυψη στο Συμβούλιο, αναφέρονται οι διάφορες αμφιλεγόμενες αρμοδιότητες. Τελικά όμως, πρέπει να πω ότι αποφάσισα με την ομάδα μου ότι θα ακολουθήσω αυτά τα οποία λέει η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι η Επιτροπή, η Επίτροπος κάνει κάποια σύγχυση με την ορολογία, διότι λέγει ότι μιλούμε για μέτρα αποκλειστικά τεχνικού χαρακτήρα από τη μια και από την άλλη λέγει ότι το όλο θέμα έχει πρακτική αλλά και πολιτική σημασία. Αυτό λοιπόν είναι εντελώς παράλογο. Απ' την άλλη πρέπει να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ και το δηλώνω ευθαρσώς ότι συμφωνώ απόλυτα με την Ισπανική Προεδρία που λέγεται ότι θα πρέπει να είμαστε λογικοί σε αυτά τα οποία κάνουμε. και εξηγούμε. Όπως είπε και ο συνάλφος Ρώμεβα και συμφωνώ μαζί του, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα ούτε οριστικό, ούτε δεσμευτικό, ούτε ουσιαστική σημασίας στην παρούσα περίπτωση. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Πρόεδρε, χωρίς να μακρηγορήσω περαιτέρω, να πω στον Μάικλ Κάσμαν ότι κατανοώ απόλυτα τους λόγους που ανέφερε και λυπούμε που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορώ να υποστηρίξω τα λεγόμενά του. Ευχαριστώ κύριε Σταβάρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι βλέπουμε ότι είμαστε μπροστά σε ένα δίλημα. Ένα δίλημα στις διάφορες πολιτικές ομάδες, προσωπικό δίλημα. Όλοι τα ίδια συναισθήματα έχουμε αυτή τη στιγμή. Ήδη πολλά μέλη εξέφρασαν τις απόψεις, η συζήτηση δεν ήταν εύκολη ούτε στις πολιτικές ομάδες, ούτε συμπεριλαμβανομένε και τι δικέ μου βεβαίω. αλλά α δούμε με σαφήνεια πού δεν υπάρχει δίλημα και πού μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι απαραίτητο στην εντολή για την Frontex να ε, δοθούν ε, κάποιες ενδείξεις για τις επιθεωρήσεις και ε, για τις διασώσεις τις οποίες κάνει στην ανοιχτή θάλασσα η Frontex. Αυτό είναι κάτι το οποίο από ανθρωπιστικής πλευράς πρέπει να το τονίσουμε και δεν θέλουμε να οπισθοχωρήσουμε, θέλουμε να προχωρήσουμε. Αντιθέτως, το συντομότερο δυνατό για να αλλάξει η εντολή της Frontex ή ε, στα πλαίσια της συναπόφασης ή όπως λέει η Άλντε σε παράρτημα. Αλλά αυτό είναι κάτι για το οποίο συμφωνούμε όλοι. Και βεβαίως θα συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε για άλλα θέματα, θα ψηφίσουμε άλλοι ναι, άλλοι όχι, αλλά μετά θα συμφωνήσουμε σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει με τον, με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο για να αλλάξει η εντολή που θα δοθεί στη φροντέρ. Εγώ ούτως ή άλλως θα υπερψηφίσω υπέρ αυτών που λέει ο κύριος Κάσμαν ε, γνωρίζοντας και τις δικές του προτάσεις, γνωρίζοντας και ποια είναι τα ε, αρμοδέντες και τα ειδικά προνόμια τα οποία έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον οποίο χαίρομαι όλοι. Θα ψηφίσω τον κύριο Κάσμαν, αλλά μετά αν θέλετε μπορούμε να προχωρήσουμε και βεβαίως κανένας δεν λέει ότι διαφωνεί ότι υπάρχουν θέματα εδώ αρνητικά. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν είναι όπως λέγουμε δεν είναι δεσμευτικά στα πλαίσια αυτών των επιχειρήσεων. Τώρα, εάν κάποιος κάνει εκβιασμό στο κοινοβούλιο, το ίδιο μπορεί να κάνει και το κοινοβούλιο στα ε, κυρίως ειδικού περιεχομένου, το ίδιο εκβιασμό μπορεί να κάνει και στα άλλα δύο θεσμικά όργανα το κοινοβούλιο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πριν από το επόμενο καλοκαίρι, αν μα πει κάποιο ότι εσεί δεν θελήσετε να κάνετε τα πράγματα όπω έπρεπε να τα κάνετε, ξέρουμε πάρα πολύ τι μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να αλλάξουμε την εντολή τη Frontex. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το όλο θέμα για να μπορέσουν όλες αυτές οι γενικές κατευθύνσεις γραμμές για την την ε, εντολή που θα δώσουμε στη Frontex να την ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό, ώστε από ανθρωπική πλευρά να μην απιστοχωρήσουμε σε αυτό που κάνουμε. Κύριε Μπουσούτιλ, γρήγορα γιατί έχουμε καθυστερήσει. Μπουσούτιλ, σύντομα ως πρόεδρε. Μας ζητείτε να εγκρίνουμε ένα μέτρο όπου ακούσαμε ότι η Κομισιόν υπερεύει τις εξουσίες της μας το είπαν αυτό είναι μικρέ υπηρεσίε, όχι μόνο μία φορά, δύο φορές μα το έχουν πει. Αν λοιπόν πούμε ναι σε αυτούς τους κανόνες σήμερα, είναι σαν να λέμε ναι σε μία περίπτωση όπου η Κομισιόν υπερεύει τις εξουσίες τη. Αυτό δεν είναι καλό σινιάλο. Βέβαια, τα περισσότερα που είχαν να υποθούν υπόθηκαν. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Απλώς ένα σχόλιο. Λυπάμαι για την πρόταση που έγινε που λέει ότι χωρί κανόνες αυτούς μερικές χώρες μέλη βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή ατόμων στη θάλασσα. Αυτό είναι η υπερβολικά πατροναριστική θέση, ιδιαίτερα για τις νότιες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Μάλτα που σώζουν ζωές στη θάλασσα εδώ και χρόνια μόνο τους. Ο ηθικό λοιπόν χάρτη που μας λέει, χαρτί μάλλον, ότι χωρίς κανόνε αυτού θα χαθούν οι είναι πολύ προσβλητικό, ιδιαίτερα για τις νότιες χώρες της Ένωσης και διαφωνώ κάθετα. Κομισιόν. Δύο λεπτά έχετε. Ευχαριστώ. Δύο σημεία. Οι γενικές αρχές και η ε, απαγόρευση ε, του μη επαναπατρισμού. Είναι απόλυτα δεσμευτικό το κείμενο, νομικά δεσμευτικό. Δεύτερον, από την πλευρά μας, οι νομικές μας υπηρεσίες, γενικώ διευθυντής, είναι διατεθειμένες να συναντήσουν την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και ενδεχομένω και του Συμβουλίου για να πάμε σε βάθος το θέμα της συζήτησης όσον αφορά την νομική διάσταση. Ευχαριστώ. Κύριε Κάσμανα, Κύριε Κορτσέτα, σας παρακαλώ. Μερικά δευτερόλεπτα έχει το λόγο Κορτσέτα. Κορτσέτα. Ήθελα να πω στον συνάδελφο Μπουζούτιλ. Εμείς ως θα αισθανόμαστε ακόμη πιο προσβελημένοι λόγω του ότι η Ιταλία, η Ελλάδα, η Μάλτα πολύ συχνά δεν βοηθάνε τα άτομα αυτά. Στη συμφωνία με τη Λιβύη έχουμε τους όρους πλήρους παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περί αυτού πρόκειται. Κάσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ λίγο την επίοικια των συντονιστών. Υπάρχει κατάργος ψηφοφορίας, δεν ξέρω, δεν έχω δει. Αν όχι, παρακαλώ η Επιτροπή μας να ψηφίσει υπέρ δηλαδή να μην αντιταχθεί στα μέτρα αυτά. Αν κάποιο δεν θέλει να αντιταχθεί στα μέτρα αυτά, πρέπει να ψηφίσει υπέρ. Αν θέλουν να αντιταχθούν στα μέτρα, πρέπει να ψηφίσουν κατά. Δεν είναι προσβολή για τις νότιες χώρες μέλη. Εγώ μίλησα για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα δύο κρατών μελών που σε 24 ώρες απέτυχαν στο να παρέμβουν και θα ήθελα αυτό να μην επαναληφθεί. Είτε περάσει αυτή η απόφαση είτε όχι. Και όλες οι απόψεις που ακούστηκαν εδώ ακούστηκαν με ειλικρίνεια και όπως είπα πριν τις σέβομαι όλους. Είμαι έτοιμος για την ψηφοφορία. Πρόεδρος. Ψηφίζουμε την πρόταση του εισηγητή. Σηκώστε το χέρι σας όσοι συμφωνείτε με την πρόταση του εισηγητή. Όσοι είστε κατά της πρότασης του εισηγητή. 25-12. Η πρόταση του συγητή απορρίπτεται. Δεύτερη ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος που ζητάει η Ολομέλεια να πάρει θέση κατά του μέτρου. Πώς είστε υπέρ του να είμαστε κατά του, του σχεδίου του μέτρου αυτού. 24. Και η κατά. Yes. Εγκρίνεται. Θα σταλεί στην Ολομέλεια. Ένα τελικό σχόλιο, κύριε Κάσπαν, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η επειδή ψήφο ήταν κατά τη σύσταση του εισηγητή, παρετούμε από εισηγητή. Εφ' λοιπόν το θέμα αυτό θα πρέπει να το φέρει στο όνομα της Επιτροπής μας ο Πρόεδρος. μάλιστα ο πρόεδρος θα το φροντίσει, η Επιτροπή μας θα αποφασίσει. Και περνάμε στο επόμενο σημείο. Colegas, por favor. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ακόμη ένα πολύ σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το 15. Σε συνδυασμό με το 14. Θα συζητήσουμε το μέλλον της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικέ υποθέσεις και το μέλλον της Eurojust μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. την Επιτροπή μας έχουμε παρόντες για τις παρουσιάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα τον Υφυπουργό για θέματα της Ισπανικής Προεδρίας, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Πρόκειται για τον υφυπουργό της Ισπανικής Κυβέρνησης κύριο Χουαν Κάρλος Κάμπο που θα μας κάνει την παρουσίαση σε σχέση με την ε, εξαιρετική όθηση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικέ υποθέσεις μας δίδει η θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα μας μιλήσει για τις ε, προοπτικές της εφαρμογής του άρθρου 86 της Νέας Συνθήκης σε σχέση με μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή για την πράσπιση των οικονομικών συμφέροντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον συντονισμό των ε, συνεργασίες των πιν, δικαστική σε θέματα ε, ποινικά διαμεθοριακό. Και μετά θα ακούσουμε και τον ε, νέο πρόεδρο της Eurojust, τον κύριο Άλετ Williams. Η Eurojust στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί και συντονίζει τον συντονισμό των, ε, της δικαστικής συνεργασίας των ε, ε, εισαγγελικών αρχών και όλων των διοκτικών αρχών σε θέματα ποινικά. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τον Υφυπουργό, μετά τον νέο πρόεδρο της Eurojust και μετά θα ανοίξουμε ζήτηση. Κύριε Υφυπουργέ, σας καλωσορίζω και δίνω μέσα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που με καλέσατε να παραστώ στην Επιτροπή σας και να σας παρουσιάσω τις ιδέες της παρούσας Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το μέλλον της δικαστικής συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει και το μέλλον τη Eurojust μετά τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Αβώνα. Σα είπα ότι με ικανοποιεί το γεγονό ότι μπορώ να λάβω το λόγο στην επιτροπή σα που χωρί υπερβολή πρέπει να σα πω ότι ενσαρκώνει το πνεύμα της νέα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσδίδουμε μεγάλη σημασία στο έργο που κάνετε και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο κύριο Λόπες Αγγιλάρ που μας κάλεσε για να ανταλλάξουμε απόψεις για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βελτιώσουμε. Σε ευχαριστούμε Χουάν λοιπόν και θα προσπαθήσουμε να είμαστε στο ύψος των με την θέση σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα την 1η Δεκεμβρίου του 2009 δόθηκε μια νέα όθηση στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Όπω γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχουν πολύ σημαντικέ επιπτώσει σε όλου του τομεί και ιδιαίτερω ε, σε σχέση με θέματα αφορούν τον πρώην τρίτο πυλώνα, ο οποίο εξασφανίζεται και σε θεσμική πλευρά είδαμε ότι σημαντικά έχουν ενισχυθεί και αυτό είναι πάρα πολύ κανονέο οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και των Εθνικών Κοινοβουλίων για τον έλεγχο της ε, ε, επικουρικότητας. Έχουμε λοιπόν ένα νέο οπλοστάσιο που βελτιώνουν τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας. Πράγμα το οποίο μας βοηθά να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και την Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μιλήσω για τους νεοτερισμούς μετά από τη ισχύει της Συνθήκης Λισαβόνα σε σχέση με τον χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης, κυρίως σε θέματα δικαστικής συνεργασίας σε ποινικέ υποθέσεις. Μετά θα αναφερθώ σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, την Eurojust και ιδιαίτερος στις προοπτικές της Eurojust για το μέλλον. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της ε, συνθήκης ο χώρος ελευθερίας δικαιοσύνης είναι ένας χώρος τον οποίο ε, ε, συμμερίζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέρη όπως εμφανίζεται στο άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη της Λισαβόνας, αν μου επιτρέπετε, αποτελεί κοινοτικοποίηση αυτού του χώρου με την γενίκευση της διαδικασίας συναπόφασης που εκ των πραγμάτων θεωρείται πλέον η συνήθις νομοθετική διαδικασία. Από δεσμικής λοιπόν άποψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 8 της συνθήκης καθορίζει τους προσανατολισμούς ε, της τραγικής που αναπτύσσεται στα πλαίσια αυτού του κοινού χώρου ελευθερίας. Το πρόγραμμα της των Χόλμης είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή όλων των αρμοδιοτήτων που δίδονται στα κράτη μέλη στα πλαίσια των αποφάσεων που λαμβάνουν και στα πλαίσια της ε, αρχής της επικουρικότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 226 ε, ε, παραμένει η νομοθετική πρωτοβουλία της Κομισιόν σε θέματα συνεργασίας, σε θέματα ποινικών υποθέσεων. Μου φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να υπογραμμίσουμε εδώ ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να μην δημιουργούμε ε, προβλήματα μεταξύ των διαφόρων ποινικών υποθέσεων, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει πραγματική συνεργασία μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών. Επίση, επιτρέπει να δοθούν νέε νομικέ βάσει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην δημιουργία αυτού του νέου χώρου ελευθερία και δικαιοσύνη. Και α, θα αναφερθώ σε αυτά τα θέματα λίγο πιο λεπτομεριακά σε λίγο. Σε σχέση με την δικαστική συνεργασία σε θέματα ποινικών υποθέσεων, το άρθρο 82 ξεπερνά τα όρια του πρώην άρθρου 31 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των ε, στόχων μιλά για την ε, ε, κατάρτιση των δικαστών και των, του υπολείπου προσωπικού των δικαστηρίων και προβλέπει διάφορα στοιχεία τα οποία αφορούν τη συνεργασία σε θέματα ε, ποινικών υποθέσεων, πάντα με συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν νέα ειδική βάση στα πλαίσια της ε, Συνθήκης Λισαβόνες που στον τομέα της ε, δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μας επιτρέπει τα εξής. Πρώτα απ' όλα, μέσω οδηγιών μπορούμε να υιοθετήσουμε ελάχιστες προδιαγραφές σε σχέση με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων. Αυτό γινόταν στο παρελθόν στον τομέα της τρομοκρατίας, της οργανωμένης εγκληματικότητας, των ναρκωτικών, αλλά τώρα και αυτές τις ελάχιστες προδιαγραφές μπορούμε να τις επεκτείνουμε στην ε, σεξουαλική ε, εκμετάλλευση γυναικών, παιδιών, ε, πλαστρογράφηση, κυβερνοέγκλημα και σε άλλους τομείς τους οποίους καθορίζει το ίδιο το Συμβούλιο. Με απόφαση ομόφωνη και με προηγούμενη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο, ανάλογα με την υπόθεση ομοφωνίας σε πλειοψηφία, καθώς και το Κοινοβούλιο, μπορεί να εγκρίνει οδηγίες για να μπορέσει να θεσπίσει τις διάφορες ε, ε, οδηγίες και κανονισμού σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του συνθήκης. Και θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι συγχρόνως με την βελτίωση της κοινή αντίδρασής μας στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία έχουμε την υποχρέωση να εναρμονίσουμε ένα ε, ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων και εγκινήσεων και διάρκεια των ε, δικαστικών ε, διαδικασιών. η συνεργασία είναι απαραίτητη και οι εγγυήσει που πρέπει να δίδουμε επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το θέμα του δικαιώματος διερμηνής και μετάφρασης και των ποινικών διαδικασιών με το οποίο ασχοληθήκατε είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό για να μπορούμε να δίδουμε τις απαραίτητες εγγύησει. Και θα πρέπει ούτως ή άλλως να προσπαθήσουμε πάνω απ' όλα να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται στο μέσο μια ποινική διαδικασίας. Κυρίες και κύριοι, εάν συμφωνούμε για τα κύρια θέματα που μας απασχολούν, να κάνουμε ταχύτερα βήματα και βήματα ποιότητος. Θα πρέπει επίσης να ε, εκθέσω με συντομία, δεδομένου ότι ο Υπουργό Δικαιοσύνη ήδη σα εξέθεσε το εξή θέμα το προηγούμενο μήνα, ότι όταν μιλούμε για δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει, οι εγγύσει είναι πολύ σημαντικέ, κυρίω για τα βήματα. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τους εγκληματίες, με την έκθεση ποινή ε, στη χώρα στην οποία κάποιος δικάζεται. Αλλά μέχρι τώρα ποτέ δεν, σχεδόν δεν έχουμε ασχοληθεί με την θέση των θυμάτων που για πάρα πολύ καιρό, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, θεωρούνταν σαν ένα απλό μέρος της όλης, ε, ε, ε, ε διαδικασίας της ποινική. Όπως ξέρετε, για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση, έχουμε μία πρωτοβουλία που, λέ που ονομάζεται ευρωπαϊκή ε, προστασία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των θυμάτων. Τα θύματα τα οποία αποτελούν θύματα οικογενειακής βίας ή βίας εξαιτίας του Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε θέματα τα οποία αφορούν τη Eurojust και το μέλλον. Με την ε, θέση σε ισχύ τη Λισαβόνα μπορούμε να εγκρίνουμε κανονισμού για να μπορέσουμε κανονίσουμε τι αρμοδιότητε τη Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 85.1 τη συνθήκη σε ισχύ. Αν και είναι δύσκολο να προσθέσω κάτι, διότι είμαι σίγουρο ότι ο Άλεντ Βίλιαμ θα σα τονίσει τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν τη Eurojust, να αναφέρω τα εξή. Η απόφαση 2002 το 86 που δημιούργησε τη Eurojust για να ενισχύεται από την ε, ε, απόφαση του Συμβουλίου Τζάι της 16 Δεκεμβρίου του 2008. Πριν από τον Ιούνιο του 2011 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την σχετική οδηγία που ε, εγγυάται τις ε, αρμοδιότητες και την εντολή της Eurojust. Οι κύριοι εταιρισμοί της απόφασης 2009 είναι η εξής. Ορισμός ενός minimum standard για τις εθνικές αρχές. Συντονισμός 24 ώρες το 23 ώρο. Δημιουργία ενός συστήματος συντονισμού με τη Eurojust. Βελτίωση των αρμοδιοτήτων του συλλογικού ε, σώματος της Eurojust και δυνατότητα να μπορέσουν να οριστούν δικαστές σύνδεσμοι σε άλλες, ε, από όλα κράτη-μέλη στη Eurojust υιοθέτηση μέτρων ε, για να γίνουν έρευνες και νέα συλλογικά ε, ε, καθήκοντα στην Eurojust, διενέργεια ερευνητικών ερευνών για να μπορέσει να ευρεθεί λύση σε περίπτωση δικαστικών διαφορών δικαστική συνεργασία όταν δεν μπορεί ένα θέμα να προσφυγεί σε δικαστική συνεργασία της Eurojust, όταν μπορεί ένα θέμα να επιληθεί μεταξύ δύο δικαιοδετικών δικαστικών οργάνων κρατών μελών. Και θα πρέπει να αναφέρω ότι τα άρθρα 85 και 86 λέγουν ότι ο ρόλος της Eurojust είναι να συνεισφέρουν στην ενήρχηση του συντονισμού των διοκτικών και ε, δικαστικών αρχών που πρέπει να συνεργαστούν δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση οικονομικών διαφορών, συντονισμός των ε, ερευνών των δικαστικών οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουμένως, δικαστική συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων ε, δικαιοδοσίας, όλα αυτά στο άρθρο 85 και στο άρθρο 86 βάσεις για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για την καταπολέμηση σε πρώτη φάση των αδικημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2001 παρουσίασε μία πράσινη βίβλο για την ε, ποινική πρόσταση των ε, οικονομικών Συμφερόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μας λέει το άρθρο 86. Ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία του είναι τα εξής. Να θεσπιστεί ότι η δημιουργία της ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής είναι πρώτα απ' όλα θέμα ευθύνης και απόβαση που θα βάλει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. η φύση αυτής της αρχής, η, ο τρόπος λειτουργίας και ό,τι αφορά την λειτουργία μιας τέτοιας αρχής είναι θέμα με των άρθρο αυτού. Εκεί αναφέρεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή σε συνεργασία με την Europol θα είναι υπεύθυνη για την αποκάλυψη αυτών οι οποίοι στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπεύθυνοι για την ε, ε, προσαγωγή τους στην ε, δικαιοσύνη καθώς και στην ανάληψη όλης της ποινική διαδικασίας για την, να τους επιβληθούν κυρώσεις. Όλα αυτά για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε εγκληματικές δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται και πέραν των συνόρων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τόσο το πρόγραμμα της οχόνομης όσο και το, πρόβλημα, ε, το πρόγραμμα των ε, τριών ε, προεδριών ασχολούνται με τα θέματα αυτά τα οποία πραγματεύονται τα άρθρα 5 και 86. Επίσης αναφέρουμε ότι μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή την τελευταία απόφαση του 2009 για να ενισχυθεί ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Eurojust και να ενισχυθούν τα καθήκοντα και οι λειτουργίες του συλλογικού της οργάνωσης. Το πρόγραμμα της ε, Ισπανικής, Βελγικής και Ουγγλικής ε, αναφέρουν ότι οι, δύο, οι τρεις προεδρίες θα αρχίσουν να σκέφτονται την ενδεχόμενη ανάπτυξη του άρθρου 86 της συνθήκες. Πράγμα το οποίο ανταποκρίνεται στο συμφέρον των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν να προχωρούν προς την οικοδόμηση του πραγματικού αυτού χώρου δικαιοσύνης και ελευθερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αρχίσει να μελετούμε το όλο αυτό θέμα για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσον μπορούμε να συστήσουμε αυτό το νέο όργανο, την νέα Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελία στην Ευρώπη κάνουμε συζητήσεις ώστε τελικά να προχωρήσουμε σε ιδέες που θα μας βοηθήσουν να ε, κάνουμε αυτή την εισαγγελία. Έγινε τον Ιούνιο του 2009 στη Μαδρίτη μια σχετική συνάντηση εμπειρογνωμόνων και πριν από κάποιους μήνες στις Βρυξέλλες έγινε μια ημερίδα με την ε, συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα της Ισπανία και ε, εκπροσώπων Τη Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής του Συμβουλίου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να συζητούν αυτά τα θέματα. Και για πρώτη φορά δόθηκε σε εκπροσώπους των κρατών μελών η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους ιδιαίτερως για αυτό το θέμα. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί, θα συνεχιστεί την επόμενη Απρίλιο, δεδομένου ότι θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο σε ένα γεύμα εργασία που θα γίνει στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνη και Εσωτερικών να συνεχιστεί η συζήτηση για αυτά τα θέματα. Έχοντας ακούσει αυτά που σας είπα, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και να αναλύσουμε όλα αυτά τα θέματα που προανέφερα για να δούμε πώς θα ενισχύσουμε και τον ρόλο της Eurojust στο μέλλον. Κατά την άποψή μας είναι πρωταρχική σημασία να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό όλες αυτές τις διαδικασίες μελέτης όλων αυτών των θεμάτων που έχουμε λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη θα πρέπει κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου μελέτη να μελετήσουμε πάρα πολύ, με πολύ σοβαρό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να συστήσουμε αυτή την ε, Γενική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να κάνουμε συζητήσεις ε, για τον, ε, τα καθήκοντά της, την εντολή της, να δούμε εάν θα πρέπει να περιοριστεί στην καταπολέμηση των ε, οικονομικών ε, εγκλημάτων στην Ευρώπη ή αν θα πρέπει να τις δώσουμε νέα καθήκοντα. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, τρεις, και, τρεις παρατηρήσεις τις οποίες θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Απλοποίηση, προσοχή, αποτελεσματικότητα. Απλοποίηση και αποτελεσματικότητα, διότι όποια και είναι η λύση την οποία θα υιοθετήσουμε, ούτως ή άλλως θα πρέπει την επικάλυψη με υπάρχοντα όργανα να την αποφύγουμε, τη στιγμή κατά την οποία κυρίως έχουμε οικονομικούς περιορισμούς παντού. Πρόκειται για μία ε, δέσμευση που αναλαμβάνουν οι δημόσιες αρχές για την προστασία των πολιτών. Αυτό το οποίο θέλουμε κυρίως να κάνουμε εμείς επίσης είναι να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όλη αυτή τη διαδικασία, όπως είπα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί δεδομένου ότι ό,τι κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε έχοντας κατά νου το πρόγραμμα της Στοχόλμης και την προστασία των πολιτών. Θέλουμε να έχουμε μια ανοιχτή Ευρώπη που να μπορεί να προστατεύει τους πολίτες της. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το κάνουμε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού χώρου Ελευθερία και δικαιοσύνη στην Ευρώπη και πιστεύουμε ότι εδώ μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο η Γενική Εισαγγελία στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που κάνατε τη σαγωγική συζήτηση για ένα θέμα τόσο σημαντικό για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης και ελευθερίας. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Γενική Εισαγγελία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό Μέχρι τώρα, όπω ξέρουμε, η Eurojust έχει παίξει πολύ, διαδραματικό ρόλο, ε, ε, πολύ ενεργητικό ρόλο σε αυτό το τομέα. Θα θέλαμε τώρα να δώσουμε το λόγο στον ε, κύριο Άλεκ Βίλιαμ, νέο πρόεδρο της Eurojust, τον οποίο συγχαίρω για την πρόσφατο ορισμό του. Έχετε το λόγο κύριε Βίλιαμς. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Δεν θα σας επιβάλλω τα ισπανικά μου. Θα μιλήσω αγγλικά μου. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να σας μιλήσω. Ο κύριος Καμπομορένο ήδη εύγλωτα παρουσίασε πολλά από τα οποία σκόπιφα κι εγώ να σας πω. Γι' αυτό θα αναφερθώ σε τρία γενικά θέματα που έχουν σημασία από τότε πάλι να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας το νέο τοπίο που έχουμε στη Eurojust η εφαρμογή το, της νέας απόφασης της Eurojust του Ιουνίου πέρυσι και το θέμα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα. Προηγουμένως δύο άλλα σχόλια. Το ένα, μετά τη Λισαβόνα, είναι σημαντική η Eurojust για την Επιτροπή σας. Διότι με τη συναπόφαση θα είστε πολύ σημαντικοί στο να δίνετε πρακτικά εργαλεία στην Eurojust για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας στην διασυνεργειακή δικαστική συνεργασία. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα συμβεί ότι θα συνεργαστούμε πλήρως. Και το δεύτερο, η αξιολόγηση που ορίζει η νέα συνθήκη να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο και για την Eurojust και για άλλα θέματα και για άλλα όργανα ποινική δικαιοσύνης. Έχουμε επίγνωση τη σημασίας αυτού του ρόλου σας. Βέβαια αυτή η αξιολόγηση ήδη ξεκίνησε. Ο διοικητικός διευθυντής μου μου είπε ότι η Επιτροπή σας είχε ήδη επαφή μαζί του σχετικά με την απαλλαγή του προπολογισμού της Eurojust. Είναι υπόλογη δηλαδή για τη δράση της ευρύτερα η Eurojust σε σχέση με τον προπολογισμό της. Και χαίρομαι για το ότι εκπρόσωπος της Επιτροπής σας θα συμμετάσχει σε μια συνάντηση τον Απρίλιο στις 20 του μηνός σχετικά με την ε, εφαρμογή της απόφασης του, της Eurojust ιδιαίτερα σε θέματα εξωτερικών σχέσεων. συμπεριλαμβανομένου και του δικαστικού ευρωπαϊκού δικτύου. Και ένα δεύτερο προεισαγωγικό σχόλιο Έχουμε, όπως σας είπα, ένα νέο τοπίο. Εγώ είμαι νεοδιοριστής. Είμαι πρόεδρος εδώ και δύο εβδομάδες μόνο. Και θα σας πω ένα ανέκδοτο, θα είναι το μοναδικό σήμερα. σε αυτά που θα σας πω μπορεί να ακούσετε πράγματα που δεν τα έχετε ακούσει, Μπορεί να ακούσετε πράγματα που είναι αληθινά, αλλά σας εγγυώμαι ότι δεν θα ακούσετε πράγματα που είναι και αληθινά και που τα ακούτε για πρώτη φορά. Για τη Eurojust λοιπόν έχουμε ένα νέο τοπίο. Σύντομα θα πάρετε την ετήσια έκθεσή μας του 2009. και θα δείτε ότι έχουμε όλο και περισσότερες περιπτώσεις που παραπέμπονται στην Eurojust από τα κράτη-μέλη για συνεργασία και συντονισμό. Το 2009 είχαμε 1.400 τέτοιες πράξεις διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας. Αύξησε 15%. Η Eurojust συναισθήθηκε το 2002. Από το 2002 μέχρι το τέλος του 2009 εφταπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις που χειρίστηκε. 1.400 περιπτώσεις πέρυσι. Εξ αυτών 130 μάλλον είχαμε 130 συναντήσεις συντονισμού που είναι η πιο πολύτιμη δουλειά μας στη Eurojust. Σε μια συνάντηση συντονισμού έχουμε εισαγγελίε, έχουμε ανακριτές από τα κρατημέλη, έρχονται στη Eurojust για να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή να προγραμματίσουν μια ημερίδα δράσης, μια καμπάνια σε σχέση με συγκεκριμένα αδικήματα ε, ευρωπαϊκό έντασμα σύλληψης να είναι έτοιμο όταν πρόκειται να γίνει μια ταυτόχρονη σύλληψη σε πάνω από μια χώρα να παγώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί εγκαίρως οι κατοίκων έρευνες να γίνουν ταυτόχρονα κλπ. έχουμε εισάγει μια νέα ταξινόμηση των περιπτώσεων. Υπάρχουν προτεραιότητες που τις ορίζει το Συμβούλιο και θέλουμε να δούμε πού είναι τα εμπόδια στη δικαστηριακή συνεργασία. Ξέρω αυτή είναι η κύρια δουλειά της Eurojust. Παίρνουμε τις προτεραιότητες του Συμβουλίου η εγκληματικότητα που δημιουργεί τα πιο πολλά προβλήματα και με αυτό τα ξυνομούμε. Τι εμπόδια τώρα συναντάμε. Αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής ε, διαπιστώσει ως εμπόδια στη δικαστική συνεργασία. Ίσως και δεν είναι έκπληξη αυτό. Είναι, προέρχονται από δύο βασικές πηγές. Η μία πηγή, πρακτική, έλλειψη πόρων και εγκληματίες εποφελούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία που έχουν και οι νομοταγείς πολίτες. Ένα παράδειγμα. Ας πούμε, έχουμε μία ομάδα εγκληματιών, συναντιόνται και βάζουν στόχο κάποιον που έχει κάνει επενδύσεις, έχει καταθέσεις και τους πείθουν να τους δώσουν τα χρήματα για άχρηστες μετοχές ή ομολογίες. Αυτό που κάνουν οι πολύ εκλεπτισμένοι εγκληματίες στην περίπτωση αυτή πάνε παίρνουν έδρα σε μία χώρα μέλος και εκεί στοχοποιούν θύματα σε άλλη, από εκεί σε άλλη χώρα μέλος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε Άγγλους κακοποιούς που σωστά από την πλευρά τους πήγαν στη Σεβίλη, στήσαν εκεί την έδρα τους, το άντρο τους. Δεν βάλαν σαν στόχο κανέναν στην Ισπανία, βάλαν σαν στόχο θύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν ξεκίνησε η ανάκριση είχαμε δυσκολίες λόγω του ότι είχαμε εγκληματίες που είχαν έδρα σε ένα κράτος μέλος και τα θύματα σε άλλο κράτος μέλος. και επειδή δεν έχουμε πολλούς πόρους αυτό ισχύει για όλες τις διοκτικές αρχές χρειάστηκε να έρθουν στην Eurojust για να λύσουν το πρόβλημα για να γίνει σωστά η ανάκριση και η συνεργασία. Για τις νομικές δυσκολίες δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τα λέει αυτά η ετήσια έκθεσή μας. Σύντομα θα την πάρετε. Μερικά είναι πολύ τεχνικά θέματα, πραγματικά για ξέπλυμα χρημάτων. Σε μερικές χώρες είναι ειδικό αδίκημα, πρέπει δηλαδή να αποδειχθεί ότι τα έσοδα από, το έγκλημα είναι αντικείμενο του ξεπλήματος. Σε άλλες χώρες το καθεστώς είναι διαφορετικό. Ο ρόλος της Eurojust είναι αυτού του είδους τα προβλήματα, καθημερινά προβλήματα στην διασυνδερική συνεργασία, να τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά. Δεύτερο θέμα, η εφαρμογή της ε, απόφασης της Eurojust και η συνάντηση του Απριλίου για την οποία σας μίλησα. Θέλαμε να κάνουμε πιο λειτουργική την Eurojust. Στο νέο αυτό τοπίο βλέπετε ότι έχουμε ένα κέντρο, τηλεφωνικό θα έλεγα κέντρο συνεργασίας που σημαίνει ανακριτές και εισαγγελείς από οποιαδήποτε χώρα μέλος μπορεί να έρθουν σε επαφή με μας οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες. 7 ε, μέρες τη βδομάδα όλο το 24ωρο. Επίσης έχουμε και υπηρεσία συντονισμού σε κάθε χώρα μέλος για να γίνει συντονισμός των πόρων, των ανθρώπινων πόρων σε κάθε χώρα και να υπάρχει και ένα άμεσο σημείο επαφής με μας. Ο Κάμπο Μορένος αναφέρθηκε στις εξουσίες της Eurojust. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, δεν θα τις επαναλάβω. Το μόνο που θα σας πω ότι λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας η υποχρέωση των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες με την Eurojust θα μας οδηγήσει μια κατάσταση όπου όταν θα έχουμε μια διασυνοριακή περίπτωση με αίτημα από μια χώρα προς δύο άλλες χώρες για δικαστική συνεργασία πρέπει να υπάρχει κοινοποίηση της περίπτωσης αυτής και στην Eurojust. Επίσης πρέπει να μας το κοινοποιούν αν υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων. Και ένα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η αυξημένη χρήση κοινών ανακριτικών ομάδων. Στο μέλλον θα είναι η πρακτική βάση συνεργασίας αστυνομίας και δικαστών. Η Eurojust μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης και αριστείας σε τέτοιου είδους κοινέ ανακριτικές ομάδες. Και ελπίζουμε να υπάρχει πια η ανάγκη των χρονοβόρων διαδικασιών μεταβίβασης επιστολών, αιτήσεων, ετοιμάτων κλπ. Και φυσικά οι σχετικές καθυστερήσεις. Όταν έχουμε μια κοινή ανακριτική ομάδα, έρχονται στην Eurojust, θα υπάρχει ειδική γραμματεία, υπάρχουν κονδύλια από την Κομισιόν, ένα παράδειγμα είναι κάτι που έγινε μεταξύ δύο κρατών μελών με στόχο περιπτώσεις εκμετάλλευσης παιδιών από το οργανωμένο έγκλημα με πολλούς τρόπους. Εκεί διαπιστώσαμε ότι για να αποσπάσουμε αποδείξεις κατά των ομάδων αυτών οι συνεντεύξεις με τα παιδιά θα έπρεπε τα παιδιά να συνοδεύονται από κάποιον και συνήθως το κατάλληλο αυτό πρόσωπο ήταν ένας συγγενής του παιδιού. Αλλά υπήρχε υποψία ο ίδιος να ήταν μέσα στο κύκλωμα που εκμεταλλεύτηκε το παιδί. Χάρη στη χρηματοδότηση αυτή νέες ανακριτικές ομάδες μπορούμε άλλοι ενήλικοι να είναι παρόντες στη συνέντευξη του παιδιού. Αυτό διευκόλυνε την αποδοχή της μαρτυρίας στο δικαστήριο μετά. Γιατί έπρεπε να είναι παρόν ένας ενήλικος στη συνέντευξη με το παιδί. Κάτι άλλο που μάλλον σας ενδιαφέρει. Σύντομα θα έχουμε και το θέμα των εξωτερικών σχέσεων που θα μας επιτρέψει να στείλουμε δικαστές συνδέσμους σε χώρες εκτός της Ένωσης. Γιατί το έγκλημα είναι παγκόσμιο. Και μέτρα πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος και εκτός της Ένωσης απαιτεί να βλέπουμε τα πράγματα ε, με έναν ε, πιο ευρύτερο τρόπο. Άρα πρέπει να υπάρξουν ανακριτές σε θέσεις και εκτός της Ένωσης. Τελειώνεται σιγά σιγά για να έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση. Δεν το έκανα οι ποιητές του Η Eurojust θέλει να συμβάλλει στη συζήτηση για τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα. Έχουμε μια ομάδα κρούσης, task force, που ασχολείται με το θέμα αυτό. Σας προσκαλούμε στη συνεδριάση της ομάδας αυτής, 28 Απριλίου παραδείγματος χάρη είναι η επόμενη. Και ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουμε με την επαγγελματική εμπειρία που έχουμε στην καταπολέμηση της απάτης στην Ένωση. Με το συλλογικό μοντέλο δράσης που έχουμε στη Eurojust και συγγνώμη αν μακρηγόρησα πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Williams. η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Χάγη, στην έδρα της Eurojust, προγραμματίστηκε με ευκαιρία την τελευταία συνάντηση των συντονιστών της Επιτροπής Λίμπες για τις 15 Απριλίου. Τότε θα επισκεφθούμε, ελπίζω, με τη Eurojust και τη Europol, ελπίζω με την ίδια μέρα, στη Χάγη. Λοιπόν, και τώρα ο λόγος στα μέλη. Έχω δει ήδη ε, κάποιους ε, συμμετέχοντες στη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους δύο προσκεκλημένους μας. Θα μιλήσω αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάμπο Μορένο. Νομίζω ότι η ομιλία σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μας και οπωσδήποτε κάθε μέλος ε, με μεγάλη χαρά θα την παραλάβει και γραπτός. Δεν ξέρω αν συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας. Δεν νομίζω ότι το Συμβούλιο θα είναι τόσο δεκτικό εις ό,τι αφορά την πρόθεση της ε, ιδέας ε, του, Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα. Αν και προσωπικά θα ήμουν ιδιαίτερα υπέρ, γιατί από τη μια είναι ε, γελίο να παραπονούμεθα συνεχώς. Βεβαίως οι εγκληματίες δεν έχουν γραφειοκρατίες, αμέσως οργανώνονται, ενώ εμάς οι αντιδράσεις μας καθυστερούν πάντα. Να συγχαρώ και τον κύριο Βίλιαμς με αυτή την ευκαιρία για την ανάληψη του αξιώματος. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις δραστηριότητες του. Ε, στηρίζω και θα στηρίζω τη Eurojust όχι μόνο γιατί ήμουν εισηγήτρια ε, για τις αλλαγές που στόχο έχουν να καταστήσουν λειτουργικότερη την Eurojust. Βεβαίως πάλι ε, έχω κάποια προβλήματα σε σχέση με το πώς αντιμετώπισε το Συμβούλιο την απόφαση πλαίσιο. Ε, επισκέπτομαι με τη Eurojust και έχω κάποιες ε, επαφές ε, πάγιες. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια αξιόπιστη υπηρεσία. Το έχει αποδείξει μέχρι τώρα και γι' αυτό δεν είμαι ιδιαίτερα ευτυχής όταν βλέπω ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν ε, κράτη-μέλη που ε, προσπαθούν να διατηρήσουν τις αρμοδιότητές τους. Κάποιες ε, σύντομες ερωτήσεις τώρα. Αναφέρατε κύριε Williams την έλλειψη πόρων σε εθνικό επίπεδο. Η ερώτησή μου είναι τι γίνεται με την έλλειψη πόρων για τη Eurojust την ίδια, γιατί Έχουμε αύξηση κατά 50, 15% ε, των υποθέσεων και μπορεί και στο μέλλον να αυξηθούν κι άλλο. Τι θα γίνει λοιπόν. Από την άλλη αναφέρεται κι άλλες δυσκολίες. Ε, νομικής φύσεως. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν νομοθετικά. Η εναρμόνιση λοιπόν σε θέματα νομικά θα βοηθούσε πολύ. Για τις κοινέ ομάδες έρευνας, εγώ είμαι υπέρ αυτών των ομάδων και δεν μπορώ παρά να διαμαρτυρηθώ, διότι ενώ το Κοινοβούλιο ψήφισε να έχετε πλήρεις αρμοδιότητες για τις ομάδες αυτές, το Συμβούλιο την τελευταία στιγμή, στο τέλος είπε ότι πρώτα πρέπει να γίνεται διαβούλευση με τα κράτη-μέλη, πριν συσταθούν οι ομάδες αυτές. Υποθέτω ότι πρέπει να χαιρετήσουμε ιδιαίτερα αυτήν την ιδέα των εισαγγελέων συνδέσμων από τη Eurojust στις άλλες χώρες, γιατί μέχρι τώρα, όπως είπαμε, ο οργανισμός αυτός απεδείχθη αξιόπιστος και ε, προστατεύει τα στάνταρ που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για την προστασία δεδομένων και για δικονομικά δικαιώματα κλπ. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βέντερ. Φαντάζομαι ότι όλοι συμμερίζεστε με τον Πρόεδρο το, την ενσυχία για την ε, έλλειψη χρόνου που έχουμε. Εμείς κανονικά θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε ε, τώρα στις 12.30 τις εργασίες μας και θα ξαναρχίζαμε στις 3. Θα ξαναρχίσουμε στις 3 δηλαδή, αλλά παρακαλούμε τους διερμηνείς να μας χαρίσουν 10 λεπτά. Και βέβαια ε, να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Ο κύριος Διαδεμέρα, χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον Υφυπουργό και να τον ευχαριστήσω για την έκθεσή του. Θα αναφερθώ στο δεύτερο μέρος, άρθρο 86, Συνθήκη της Λισαβόνας. Μας είπε ότι η δημιουργία της εισαγγελία αυτής θα πρέπει να έχει κύρια χαρακτηριστικά τρία. Ε, ομοφωνία, πρώτερη συμφωνία του Κοινοβουλίου, δεν μας είπε για την τρίτη. Όταν δεν υπάρχει ομοφωνία, μιλάμε για ενισχυμένη συνεργασία. Αν δεν υπάρχει ομοφωνία, όμως πώς βλέπετε να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία. Δεύτερη ερώτηση για τον κύριο Βίλιαμ, τον οποίο θέλω να συγχαρώ πρώτα απ' όλα. Όταν ήταν εδώ ο κύριος Λόπης Μότα μας σκανδάλισε όταν είπε ότι δεν έχουν κύριες πηγές πληροφόρησης και το 80% προέρχονται από τα ΜΜΕ. Αυτό είναι δραματικό. Δεύτερη ερώτηση. Δεν σας άκουσα να μιλάτε για ανταλλαγή στοιχείων από τα ποινικά μητρώα για να διευκολύνετε την κατάστασή σας όταν έχετε να κάνετε με εγκληματίες. Μιλήσατε για κοινέ ε, ερευνητικές ομάδες, για ανακριτικές ενώ πιο προσεκτική η Ισπανική Προεδρία μιλάει για κοινέ ομάδες ε, συνεργασίας. Παρακαλώ λοιπόν αυτή την αποχρώσα διαφθορά να μου την ε, ε αναλύσετε. Ο κύριος Χάρογκη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την καταδίκη μου για την δολοφονία ενός αστυνομικού από ένα μέλος της ΕΤΑ. Οι δύο ερωτήσεις για τους δύο εισηγητές. Κύριε Κάμπο που είναι το πακέτο διαδικαστικών μέτρων που διαθέτουμε για τις ποινικέ διαδικασίες στην Ευρώπη. Η μετάφραση είναι ένα στοιχείο, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Πολλές άλλες οδηγίες και κανόνες που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ εγκληματολογικών αρχών για την Ισπανική Προεδρία στα πλαίσια του προγράμματος της Στοχόλμης. Πού βρίσκεται το πακέτο των μέτρων για τις εγγύησεις κατά τη διάρκεια της ποινική διαδικασίας. Διότι καλό είναι να μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον Εισαγγελέα, αλλά φοβούμε ότι δεν θα ξεπεράσουμε κατά πολύ το στάδιο των συζητήσεων που θα γίνει στο Συμβούλιο και με την κυρία Βέμπερ συμμερίζουμε την ιδέα ότι δυστυχώς για το θέμα αυτό είμαστε ακόμη πολύ μακριά. Καλό θα είναι λοιπόν να εκθέτει το θέμα η Ισπανική Προεδρία και ίσως κατά τη διάρκεια του επιδορπίου να ανταλλάσσει και κάποιες απόψεις. Αλλά, δεν, αλλά νομίζω ότι από μη πόρο απέχουμε από την υλοποίηση αυτής της ιδέας. Κύριε Βίλιαμς, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πιστεύετε ότι η εθνική εκπροσώπηση στην Eurojust είναι αποτελεσματική, είναι επαρκής, είναι σταθερής ο τρόπος τον οποίο συνεργάζονται τα κράτη-μέλη, διότι αυτή είναι η εντύπωση που μας έδωσε και στον κύριο Ντίεφ Δεμέρα και σε μένα η προηγούμενη παρουσίαση που έκανε ο κύριος Μότα, ότι η συνεργασία η εθνική δεν είναι επαρκής. Η θεσμική παρουσία δεν είναι η καταλληλότερη στη Eurozone, δηλαδή ότι δεν είναι σταθερή και αποτελεσματική η εθνική εκπροσώπηση. Ευχαριστώ. Για τους συναδέλφους που έφτασαν ε, αργά και για τον κύριο Υφυπουργό θα ήθελα να σας πω ότι εγώ άρχισα τη συνεδρίαση καταδικάζοντας ε, ε ρητά την ε, τρομοκρατική αυτή ενέργεια της ΕΤΑ, την δολοφονία του Γάλλου αστυνομικού και εξέφρασα την αλληλεγγύη μου προς την οικογένεια του θύματος και την αλληλεγγύη όλων μας σε θέματα κατά πολέμης τρομοκρατίας. Κυρία Ρωσελίνο. Σας ευχαριστώ για τα πολύ ε, σαφή και ακριβή που μας είπατε και συγχαρητήρια στην κυρία Βίλιαμς για το διορισμό του. Εγώ ξεκινάω από τη δική μου εμπειρία. Εγώ με από τη Σικελία και δυστυχώς έζησα και ζω δύσκολες καταστάσεις. Ευχαριστώ την προσοχή σας σε δύο προβλήματα που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα τύπου μαφία. Το ξέρετε καλύτερα από μένα πόσο διαφορετική είναι από το οργανωμένο έγκλημα γενικότερα. Έχει δύο μορφία η μαφία. Δύο λοιπόν. Το ένα αναφερθήκατε στην προστασία των θυμάτων, η προστασία των μαρτύρων και προστασία ζωής και ποιότητα ζωής. Συχνά ξεριζώνονται τα άτομα αυτά από το χώρο που ζούσανε, από τη ζωή τους την ίδια και ζούνε σε δύσκολες συνθήκες. Και το δεύτερο, η κατάσχεση της περιουσίας, της μαφίας, που είναι ένα όργανο που εφαρμόζεται, χρησιμοποιείται στην Ιταλία. Πολύ σημαντικό θα ήταν να επεκταθεί για την Ευρώπη, γιατί η μαφία έχει διεθνοποιηθεί, ξεπερνάει τα σύνορα πια. Τα περιουσία, οι επενδύσεις των μαφιόζων σίγουρα υπάρχουν σε κάθε χώρα. Στην Ιταλία επιπλέον έχουμε ένα νόμο που επιτρέπει την κοινωνική χρήση των, της κατασχεμένης αυτής περιουσίας που είναι σημαντικό και οικονομικά και ως μήνυμα προς τους εγκληματίες και προς τους πολίτες και επηρεάζει φυσικά και την παρουσία των μαρτύρων. Τα δύο θέματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Κύριε Κολίνο. θα είμαι πολύ σύντομος. Εύχομαι καλή δουλειά και στον κύριο Μαρένο και στον κύριο Βίλιαμ. Σε ερώτηση. Πρόσφατα με μια αντιπροσωπεία πήγαμε στην Καλαβρία και στη Ρώμη. για την κοινωνική προστασία των εργαζομένων από τρίτες χώρες το θέμα. Στη Ρώμη συναντήσαμε τον Γενικό Εισαγγελέα για θέματα μαφίας και τους συνεργάτες του. Συζητήσαμε και σας παρουσιάζω μερικά σχόλια από τη συνάντηση αυτή. Δύο συγκεκριμένα προβλήματα. με ό,τι μορφή και να παίρνει το οργανωμένο έγκλημα και για όποια χώρα να πρόκειται. Πρώτη δυσκολία, οι κατασχέσεις είναι δύσκολες. Βέβαια, συζητήσαμε για την Ιταλία, αλλά υπάρχουν δυσκολίες ανάμεσα στο κράτος που παίρνει την απόφαση της κατάσχεσης και το κράτος που πρέπει να το εκτελέσει. άλλο θέμα κάτι που τον άφησε στον Γκράσο είναι πολλές χώρες ακόμα σήμερα αρνούνται την ύπαρξη της μαφίας ή του οργανωμένου εγκλήματος στον χώρο τους, στο εδεφός τους. Λένε ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά άλλες χώρες. Και διερωτώ με. Άρθρο 86 αν οριστεί αυτός ο εισαγγελέα κατά της μαφίας υπάρχουν όρες συγκεκριμένοι που θα μας επιτρέψουν να οργανωθούν οι δραστηριότητες τους 1400 περιπτώσεις συνεργασίας είπατε αλλά ο πολίτης κυρίως έχει συνδέσει τη Eurojust με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εύχομαι μέσα αυτή εδώ την πενταετία από κοινού να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ο επόμενος συνάδελφος. Ο κύριος Κάμπος μίλησε για ελάχιστα πρότυπα εγκλημάτων και ποινών. Τι εννοούσε ακριβώς. Το περιορίζει σε εγκλήματα διασυνοριακά όπου υπάρχουν παράλληλοι ορισμοί, αν γίνεται στα κράτη-μέλη το έγκλημα ή στα σύνορα ή εναρμονίζεται ο ορισμός όλων των διασυνοριακών εγκλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βέβαια τα τρία διακριτά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου θα ε, υπονομευθούν. Ε, δηλαδή, ε, τι ακριβώς εννοείται με αυτό που είπατε, ότι θα υπάρξει αλλαγή και σε σχέση με τα συστήματα που υπάρχουν στην Αγγλία-Ουαλία. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε τώρα πρώτα τον κύριο Βίλιαμς και μετά τον κύριο Υφυπουργό. Κύριε Βίλιαμς, ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν θα απαντήσω με τη σειρά. Θα απαντήσω πρώτα στον κύριο Χάριγκη και την εκπροσώπηση της στη Eurojust. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η νέα απόφαση για τη Eurojust θα απαιτεί από τα κράτη-μέλη να έχουν όχι μόνο εθνικό αντιπρόσωπο, αλλά και βοηθούς και αναπληρωτές. Ελπίζομαι ότι αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη κάλυψη των επιχειρησιακών μας δραστηριοτήτων. Τώρα, η κυρία Βέντερ ε, Βεβαίω, υπάρχουν ε, δημοσιονομικά προβλήματα. Ο προπολογισμό συνεχίζει να μας απασχολεί. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη που ε, την αναγνώρισε να δούμε πέρα από τα μέσα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουμε συνεργασίες με τις δικαστικές αρχές. Ο κύριος αναφέρθηκε στις πηγές πληροφόρησης της Eurojust. Θα ήθελα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο και να θέσω το ζήτημα της πρόσβασης σε αρχεία Μητρώα. Σε ό,τι αφορά το πιο στενό θέμα της πρόσβασης σε Μητρώα, αυτό είναι ένα αίτημα στα πλαίσια της νέας απόφασης της Eurojust ότι τα εθνικά μέλη και οι βοηθοί τους στην Eurojust θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μητρώα, καταδίκες κλπ. κοινικά μητρώα κλπ. Τώρα, γενικότερα, εις ό,τι αφορά το θέμα των πηγών, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Eurojust χρησιμοποίησε σε στενή ε, συνεργασία με τη Europol, και αυτό είναι σημαντικό, ε, ε, μια υπηρεσία επεξεργασίας πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή συστεγαζόμαστε στη Χάγη και επειδή έχουμε στενές σχέσεις με την ε, Europol, έχουμε πρόσβαση μέσω της Europol σε ε, πληροφορίες. Το άλλο θέμα που έθεσε ο κ. Δίας Δεμέρα είναι η διαφορά μεταξύ κοινών ερευνητικών ή ανακριτικών ομάδων και ε, μεικτών ομάδων συνεργασίας. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ευνηδιάστηκα λίγο γιατί δεν ήξερα ότι στην Ισπανία γίνεται αυτή η διάκριση. Σε ό,τι αφορά τη Eurojust, εμείς έχουμε ένα εγχειρίδιο για τις κοινέ ανακριτικές ομάδες και θεωρούμε μια κοινή ανακριτική ομάδα ή κοινή ερευνητική ομάδα ως μια ομάδα που σκοπό έχει μεταξύ άλλων να διευκολύνει την συνεργασία και το συντονισμό των ενεργειών μεταξύ εθνικών αρχών. Ε, ο κύριος Γιακολίνο και η κυρία Μπορσελίνο. Τώρα, βεβαίως, ε, έχουμε επίγνωση του, της σημασίας του θέματος των κατασχέσεων ε, κλπ. Επί Ισπανικής Προεδρίας η Eurojust θα οργανώσει ένα σεμινάριο για αυτό το θέμα. Δυσκολίες δηλαδή ε, κατασχέσεων ε, προϊόντων ξεπλήματος χρημάτων. Ε, οι υπόλοιπες ερωτήσεις νομίζω ότι αφορούν τον κύριο Κάμπο Μορένο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους σας για τις, ε, τα συγκεκριμένα σχόλιά σας Συμφωνώ και εγώ με την υποστήριξη των θυμάτων και την τρομοκρατική ενέργεια τη χθεσινή. Με τα εργαλεία που έχουμε μπορούμε να ξεριζώσουμε αυτή την τρομοκρατία από τις χώρες μας. Πολλές ερωτήσεις έγιναν. Θα ήθελα να τις απαντήσω όλες με τη σειρά, με παιδαγωγικό τρόπο. Φυσικά αυτό έχει σχέση με την παρέμβασή μου στην αρχή. Όντως είμαι αισιόδοξο. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, διότι έχουμε τα νομικά μέσα που μας επιτρέπουν να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να κάνουμε δηλαδή μια ισχυρή Ευρώπη που θα μπορεί να είναι στην υπηρεσία των θυμάτων, να ακούει τι έχουν να πούν τα θύματα. Έχουμε ήδη το προσχέδιο αυτής της νέας Ευρώπης που θέλουμε να κάνουμε και προσπάθησα εγώ να σας ε, εξηγήσω, να σκιαγραφίσω μάλλον ποιες είναι στον τομέα αυτό που μας απασχολεί τα σχέδια της Ισπανικής Προεδρίας. Σας έλεγα ότι ξεκινούμε από την ανάγκη και από αυτά που μας προσφέρει το άρθρο 86 καθώς και από νέα πράγματα. Βεβαίως πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό και κύριε Διαδεμέρα στην δεύτερη και τρίτη παράγραφο προβλέπεται τι γίνεται σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί η ομοφωνία. Επιμένω όμως. Δεν είναι σήμερα η συγκεκριμένη κρυμενοποίηση του προτύπου που μας απασχολεί. Απλώς πρέπει να αρχίσουμε κάποια στιγμή και το κάποια στιγμή είναι σήμερα. Ας αρχίσουμε σίγουρα και, σήμερα και θα προχωρήσουμε σίγουρα. Και αν δεν αρχίσουμε να κάνουμε σημαντικά βήματα προς τη δημιουργία μηχανισμών που θα μας επιτρέψουν να εκριζώσουμε γενικά, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται ένας προοδευτικός μηχανισμός στην συνθήκη, αν δεν αρχίσουμε σήμερα, αν δεν αρχίσουμε σήμερα λοιπόν να κάνουμε κάτι για να δημιουργήσουμε αυτή τη γενική εισαγγελία κατά των οικονομικών εγκλημάτων στην Ευρώπη, δεν κάνουμε τίποτα. Σημαίνει αυτό ότι επικρίνουμε την Όλαφ ή την Eurojust. Όχι. Απλώς λέμε ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πιο δυναμικούς, πιο ισχυρούς μηχανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε ε, σήμερα να καταπολεμήσουμε αυτή τη μορφή της οργανωμένης εγκληματικότητας. Εάν 21ος αιώνας θεωρείται ότι ο χρυσός αιώνας της οργανωμένης εγκληματικότητας, θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Και σήμερα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε όχι ο καθένας χωριστά, αλλά ως οργανωμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να μπορέσει να δημιουργήσει τους μηχανισμούς που σε συνεργασία και σε συντονισμό με την διεθνή κοινότητα και τα κράτη-μέλη να μπορέσει να εκριζώσει αυτές τις εγκληματικές πρακτικές πολλές ε, φορές ε, ε, προέρχονται και από την αποδυνάμιση των εθνικών συνόρων. Σήμερα όμως πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση αυτή και όχι αύριο. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα για αύριο και θα πρέπει να κάνουμε τα διάφορα βήματα που πρέπει να κάνουμε το συντομότερο δυνατό. Και γι' αυτό σας μίλησα για τρεις προτεραιότητες, τις οποίες ούτως ή άλλως η αναζήτηση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και η ιδιαίτερη προσοχή που θα δώσουμε σε όλες τις δράσεις που θα αναλάβουμε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε σήμερα. Και ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος, αλλά είναι ανάγκη να κάνουμε με τα μέσα τα οποία θα δημιουργήσουμε μια πιο ισχυρή Ευρώπη, για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την, σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μπορούν να ζουν οι σημερινές τους κοινωνίες πιο ήσυχοι. Ευχαριστώ. Ραμόν Χάουραγγι. Προχωρούμε. Προχωρούμε στο θέμα των εγγύσεων για τις ε, δικαστικές διαδικασίες. Ίσως ε, πιο γρήγορα από ό,τι μας αφήνουν να βλέπουμε τα γεγονότα. Έχουμε με ένα φύλλο πορείας, ένα χάρτη πορείας, ο οποίος έχει σκεγγραφηθεί πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θα πρέπει όμως να περιοριστούμε στα λόγια, πρέπει να προχωρήσουμε με έργα και να κάνουμε βήματα προοδευτικά. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν αυτά τα βήματα ξεκινώντας από κάπου. Το πρώτο βήμα, είπαμε, είναι για την προστασία όλων η μετάφραση και διερμηνία και διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Όταν ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα θα περάσουμε στο δεύτερο. Αλλά ούτως ή άλλως θα πρέπει σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες να εξασφαλίσουμε έναν κοινό παρανομαστή. Διότι οι εγγύσεις είναι πολύ σημαντικές και οι εγγύσεις θα πρέπει σε όλες τις χώρες να δίνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους πολίτες. Και βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε ε, και εθνικό επίπεδο, αλλά κυρίω να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα όσον αφορά τις εγγύσεις τις οποίες δίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να δώσουμε τις εγγυήσεις που χρειάζεται να δώσουμε σε όλα τα θύματα και σε όλους τους πολίτες που τη χρειάζονται. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να δώσουμε μία, ένα πάρα πολύ ε, σημαντικό βήμα προς τα μπρος για να ικανοποιήσουμε τον πρώτο στόχο της, ε, του χάρτη πορείας και μετά αφού μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πρώτη πρόκληση να προχωρήσουμε στη δεύτερη. Κάπου πρέπει να αρχίσουμε και πρέπει να αρχίσουμε γρήγορα. Αυτή είναι μια νέα ιδέα, μια νέα ανάγκη. Έχουμε όμως την δυνατότητα να έχουμε ένα μηχανισμό ισχυρό στη διάθεσή μας και αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε την Ευρώπη πρέπει να σταματήσουμε τις ε, άχρηστες και αέναες συζητήσεις, να σηκώσουμε τα μανίκια και να αρχίσουμε τη σκληρή δουλειά από κοινού. Κυρία Μπορσολίνο, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην Ισπανία. Έχουμε κάνει επίσης ε, ε, πολλές συζητήσεις για να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα των λαθρεμπορίων ναρκωτικών που μας απασχολεί όλους ιδιαίτερως και εμάς όπως και τη χώρα σας. Και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό χωρίς να, μπορέ, χωρίς να χρειαστεί να εξαντλήσουμε τις πηγές που έχουμε. Και βεβαίως στην ε, η μερίδα που θα οργανώσουμε τον Μάιο θα ασχοληθούμε με όλα αυτά τα θέματα ώστε να σταματήσουμε και την παράνομη ε, κυκλοφορία κεφαλαίων, να σταματήσουμε το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, το οποίο κάποια στιγμή δηλητηριάζει τη ζωή όλων μας. Ελπίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τελειώνω σε μια Ευρώπη ισχυρή, μια Ευρώπη που θα αισθάνεται ασφαλής και στα πλαίσια της λειτουργίας μας με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να έχουμε μια νέα Ευρώπη που θα ζει ακόμη πιο ειρηνικά. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για τους διερμηνείς που μας χάρισαν ακόμη ένα τέταρτο και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, προσκεκλισμένους μας παρέστησαν στις ε, συζητήσεις. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υφυπουργό, τον ε, κύριο Williams, νέο πρόεδρο της Eurogest. Διακόπτουμε και θα συνεχίσουμε σήμερα το απόγευμα στις 3.